Bene, riprendiamo il lavoro. Πολύ καλά και αρχίζουμε και πάλι τις εργασίες μας για τις νέες ευκαιρίες για τα δύο φύλλα μετά το 2015. Ξεκινάμε βέβαια ορισμένοι συνάδελφοι έρχονται τώρα αλλά δεν μπορούν να καθυστερήσουν πολύ μετά από την κανονική ώρα οι διερμηνείς, γι' αυτό θα πρέπει να βιαστούμε. Θα πρέπει να ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος του σεμιναρίου αυτού, γιατί ε, διέρχησαν παραπάνω σήμερα το πρωί και ε, μέχρι τις 3.30 θα είμαστε με την ε, ειδική εισηγήτρια και θα έχουμε επίσης ερωτήσεις μετά που θα υποβληθούν και θα μας απαντήσει. Ντρότα Σέλεβα με, από το Πανεπιστήμιο της ε, Βαρσοβίας και με πιστή και θα μας μιλήσει για την μητρική άδεια, την άδεια Η Δροτά έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τους οργανωτές για την πρόσκληση που μου απίθυναν. Χαίρομαι ιδιαίτερως που βρίσκομαι εδώ. Το καθήκον που μου ανατέθηκε είναι να κάνω μια αναθεώρηση των δράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την άδεια μητρότητας και την άδεια πατρότητας. Να προσπαθήσω να τις αξιολογήσω και να καταλήξω σε ορισμένες συστάσεις. Είναι πολύ ευρύ το πεδίο αυτό και νομίζω ότι μπορέσαμε να κάνουμε μια πολύ σωστή επισκόπηση της εργασιακής κατάστασης γυναικών και ανδρών κατά τη διάρκεια της πρωινής μας συνεδρίασης και τέθηκαν διάφορα προβλήματα σε σχέση με τα γυναικεία ποσοστά απασχόλησης. Και τα αναφέρω αυτά τα βασικά προβλήματα γιατί έχουν άμεση σχέση με την εξισορρόπηση εργασιακής και οικογενειακής ζωής, με τη συμφιλίωση της εργασίας και της οικογένειας και τα προβλήματα που εγείρονται με την άδεια μητρότητας και πατρότητας, διότι αυτά αποτελούν μέρος του προηγούμενου προβλήματος που σας ανέφερα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τις τελευταίες δύο δεκαετίες παρατηρούμε το εξής, τα ποσοστά γυναικείας απασχόλησης αυξάνονται. Ωστόσο, μένει το χάσμα μεταξύ των δύο φύλων στο χώρο εργασίας. Υπάρχει ας πούμε μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων και διαφορές ε, εντοπίζονται μεταξύ κρατών μελών ως προς το πώς αυξάνεται το ρυθμό αύξησης του ποσοστού απασχόλησης των γυναικών και μάλιστα σε χώρες του Νότου της Ευρώπης και σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης ε, η ανεργία των γυναικών είναι πολύ μεγαλύτερη και αυτό το πρόβλημα είναι πολύ οξύ. Κάτι το οποίο αναμένεται να οξυνθεί και στο μέλλον και να θέσει σε κίνδυνο την οικονομική τους κατάσταση αλλά και την αυτονομία τους. Και υπάρχουν και διαφορές μεταξύ των διαφόρων ηλικιακών ομάδων. Εάν δούμε τους δείκτες της, ε, των ποσοστών γυναικείας απασχόλησης βλέπουμε ότι αυξάνεται η απασχόληση των γυναικών σε ε, μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες, αλλά η αύξηση της απασχόλησης των νέων γυναικών δεν είναι τόσο σημαντική. Ε, ακόμα στην Ευρώπη λοιπόν παρατηρούμε αυτό το οποίο αποκαλούμε το την ποινή της μητρότητας. Δηλαδή η απασχόληση των ε, γυναικών που έχουν παιδιά είναι πολύ μικρότερη των γυναικών που δεν έχουν παιδιά ή που δεν, τα, ε, δεν είναι οι μόνες που είναι επιφορτισμένες με, την, ε, με το μεγάλωμα και την ανατροφή τους. Όταν αυτά είναι σε πολύ μικρή ηλικία βεβαίως. Και γι' αυτό έχουμε διάφορες δράσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και εθνικές πολιτικές που αποσκοπούν στην καταπολέμηση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των δύο φύλων και στην εξάλληψη της, του πέναλτη, αν θέλετε, με την ποδοσφαιρική έννοια του όρου, της ποινή δηλαδή που υποχρεώται να, καταλάβει, να καταβάλει η γυναίκα για το ότι γίνεται μητέρα. Η άδεια μητρότητας και η άδεια πατρότητας δίδονται συνήθως αμέσως μετά το κετό. Είναι σημαντικό για τη γυναίκα να ανακτήσει τις δυνάμεις της μετά τον τοκετό, να μπορέσει να εδραιώσει τον θυλασμό. Αυτές είναι πολύ σημαντικές περίοδοι της ζωής ενός ζευγαριού και θα πρέπει να αλλάξει η διοργάνωση του νοικοκυριού, ο τρόπος με τον οποίο γίνονται τα πράγματα σε κάθε οικογένεια και για τους πατερές είναι σημαντικό αυτό να μπορέσουν να έχουν άδεια πατρότητας για να αναπτύξουν γονεϊκές δεξιότητες και να αναπτύξουν δεσμό με το νεογέννητο παιδί τους. Η οδηγία λοιπόν θέτει ένα πρότυπο 14 εβδομάδων για την άδεια μητρότητας και φαίνεται αυτό ξεπερασμένο εν ώψη μάλιστα του γεγονότος ότι στα περισσότερα αν όχι σε όλα τα κράτη-μέλη ήδη τηρείται αυτό, αυτή η νόρμα, αυτό το ελάχιστο πρότυπο και μάλιστα σε νομοθεσίες ορισμένων χωρών και μάλιστα πολλών χωρών βλέπουμε ότι είναι πολύ υψηλότερα και καλύτερα τα πρότυπα που προβλέπονται, τουλάχιστον 18 εβδομάδες ε, πληρωμένης άδεια μητρότητας π.χ. στα κράτη-μέλη της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Ως προς την άδεια πατρότητας, δεν υπάρχει πρότυπο αυτή τη στιγμή σε ευρωπαϊκό επίπεδο, απλά έχει ε, χαρακτηριστεί αυτό, έχει σημανθεί ως ανάγκη δεν υπάρχει ενιαίο πρότυπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση για άδεια πατρότητας που μπορεί να πάρει ένας πατέρας αμέσως μετά τη γέννηση του παιδιού του. Ε, δεν υπάρχει ένα ευρωπαϊκό πρότυπο, έχουμε μια πλειάδα διαφορετικών λύσεων αναχώρα μέλος. Σε αυτή τη μελέτη και σίγουρα ε, την είδατε το πρωί γιατί ήταν στην, ε, στην αίθουσα, στην είσοδο της αίθουσα κατά την πρωινή συνεδρίαση, έχουμε εκεί ένα συγκριτικό πίνακα που δείχνει ότι τα κράτη-μέλη προσπαθούν να δώσουν τέτοιες λύσεις με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους για τις μητέρες και τους πατέρες της εκάστοτε χώρες. Ωστόσο, αυτό το οποίο είναι σύνηθες είναι και το εξής. Στην πλειονότητα των χωρών η γυναίκα είναι αυτή που αποφασίζει να ε, πάρει την α, γονική άδεια, την άδεια μητρότητας. Όταν αυτή τελειώνει, ε, ο εργαζόμενος ε, παίρνει γονεϊκή άδεια, άδεια γονέων. Αξιοποιεί δηλαδή άλλες δυνατότητες να απουσιάσει. Αυτή η άδεια συνήθως διατίθεται και στους δύο γονείς, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις δεν μπορεί να μεταφέρεται και αποτελεί ατομικό δικαίωμα του ενός γονέα. Οι έρευνες δείχνουν το επεργέτημα της άδειας γονέα. Εάν η περίοδος αυτή είναι εξαιρετικά μεγάλη, βλέπουμε ότι μπορεί να αυξήσει την ποινή που καταβάλει μια εργαζόμενη γυναίκα για το ότι γίνεται μητέρα. Δηλαδή η, μακριά, η μεγάλη απουσία από το χώρο εργασίας την κάνει να δυσκολεύεται να επανέλθει στο σημείο που βρισκόταν και θα έχει μικρότερες ανταμοιβέ. Υπάρχει κάτι το ευεργετικό, αλλά υπάρχουν και αρνητικές επιπτώσεις. Ωστόσο, το πιο σημαντικό ε, εδώ είναι το εξής. Οι πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να εμπλακούν οι πατέρες στη φροντίδα των παιδιών. Και είναι ένα εργαλείο άσκησης πολιτικής αυτό, το οποίο ε, μπορεί να επηρεάσει τη συμπεριφορά και να την αλλάξει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Έχουμε λοιπόν την οδηγία για την γονική άδεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όμως ο ελάχιστος κοινό παρονομαστής είναι πραγματικά πολύ, πολύ μικρός. Υποχρεώνονται τα κράτη-μέλη να παρέχουν τουλάχιστον τέσσερις μήνες και λέει η οδηγία ότι τον ένα μήνα θα πρέπει οπωσδήποτε να τον πάρει ο ένας από τους δύο γονείς. Ότι ο κάθε γονιός πρέπει να πάρει τουλάχιστον τον έναν από τους τέσσερις. Και ε, δεν ε, το δέχονται πολύ αυτό όταν δεν έχουν επαρκή ανταμοιβή για την σημασμένη περίοδο, για την περίοδο που έχει τεθεί κατά μέρο έτσι ώστε να απουσιάσει ο εργαζόμενος. Μάλιστα, στις χώρες όπου η άδεια πατρότητα συνοδεύεται από, από ε, ευεργετήματα, από επιδόματα, τότε μόνο ο πατέρας ε, ε, κατά πάσα πιθανότητα επιλέγει πράγματι να πάρει αυτή την άδεια. Εάν δεν συνοδεύεται από κάποιο επίδομα, σπάνια ή και καθόλου ο πατέρας επιλέγει να απουσιάσει από την εργασία του. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλες λύσεις. που αποσκοπούν να βοηθήσουν τις οικογένειες να συμφιλιώσουν την εργασιακή με την οικογενειακή τους ζωή. Δηλαδή ευέλικτος χρόνος εργασίας, ευέλικτο ωράριο, ε, μια μεταβατική περίοδος όταν οι γονείς επιστρέφουν στη δουλειά είναι κάτι το οποίο γίνεται σε συνεργασία ενδεχομένω με τον εργοδότη και θα πρέπει να γίνεται έτσι για να υπάρξουν διάφορες διευθετήσεις για να προσαρμοστεί ο χρόνος εργασίας στις ανάγκες μιας οικογένειας η οποία έχει ε, παιδί. Ωστόσο, και πάλι, κυρίως γυναίκες επιλέγουν αυτή την άγωσα Και οι ρυθμίσεις αυτές πολύ συχνά είναι συνδεδεμένες με χαμηλότερο μισθό, με, με μειωμένες ώρες εργασίας. Και άρα αυτό συμβάλλει στο μισθολογικό χάσμα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ορισμένες φορές βεβαίως είναι καλύτερο για τις ε, μητέρες και τους πατέρες να μειώσουν το ωράριό τους, ωστόσο οι γυναίκες είναι αυτές οι οποίες κατά κύριο λόγο επιλέγουν αυτή τη ρύθμιση και άρα εργάζονται λιγότερες ώρες, κερδίζουν λιγότερα χρήματα και πάλι υφίστανται αυτή την ποινή της μητρότητας. Για αυτόν ακριβώς το λόγο. Τέλος, πέρα από τα εργαλεία πολιτικής που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, τις ε, οικογενειακές άδειες, Υπάρχουν και οι υπηρεσίες φροντίδας των παιδιών. Θεσμικά δηλαδή ε, προσφέρονται ε, υπηρεσίες φύλαξης μέρημνας φροντίδας των παιδιών. Το πιο γνωστό εργαλείο συντονισμού τέτοιου είδους πολιτικών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι οι γνωστοί στόχοι της Βαρκελόνης, οι, οποίες τέθηκα, οι οποίοι τέθηκαν το 2002. Μέχρι σήμερα μόνο 9 χώρες συμμορφούνται με τον πρώτο στόχο που είναι το 33% των παιδιών από 0 ως 3 ετών να έχουν μπει σε τέτοιες δομές. Και περίπου 50 ε, είναι το ποσοστό των παιδιών που προσχωρούν σε τέτοιες δομές ε, φροντίδας από, στην ηλικιακή ομάδα των 3 έως 6 ετών. Και βλέπετε ότι οι χώρες που εκπληρώνουν τους στόχους της Βαρκελόνης για τα παιδιά κάτω των 3 ετών είναι και οι χώρες που παραδοσιακά και ανέκαθεν αν θέλετε είχαν υψηλή πρόσβαση, παρήχαν μεγάλη πρόσβαση σε τέτοιου είδους υπηρεσίες. Και είναι βεβαίως οι ίδιες χώρες που εκπληρώνουν και το δεύτερο στόχο της Βαρκελόνης ως προς τους παιδικούς σταθμούς και τα νηπιαγωγεία. Και Υπάρχουν και νέες ανάγκες της οικογένειας, εκτός από τη φροντίδα των παιδιών στο πλαίσιο της γύρανσης των κοινωνιών μας. Έχουμε τη γενιά σάντουιτς, έτσι την αποκαλούμε. Γυναίκες 60 ετών, οι οποίες συνεχίζουν να είναι δραστήριες επαγγελματικά, έχουν όμως μεγαλύτερους σε ηλικία γονείς, τους οποίους ε, πρέπει να φροντίζουν και έχουν και εγγόνια τα οποία πρέπει να φροντίζουν. Αναμένεται από αυτές να φροντίζουν τους υπέργυρους γονείς, της, γονείς τους, να ε, φροντίζουν τα εγγόνια τους και να συνεχίζουν να είναι δραστήριες επαγγελματικά επίσης. Νέες είναι οι προκλήσεις που υψώνονται επομένω ε, στον τομέα της μακροπρόθεσμης περίθαλψης ή φροντίδας και έχει σημασία να τα συζητήσουμε όλα αυτά όχι μόνο στο πλαίσιο της συζήτησης για τη φροντίδα των παιδιών. Τέλος, στη μελέτη μας δίδουμε μία σειρά συστάσεις. Μία σειρά συστάσεων για τις ε, γονικές άδειε και για τη θεσμική, θεσμικώς κατοχυρωμένη φροντίδα των παιδιών. Θα αναφερθώ εν συντομία. Είναι σημαντικό να αναθεωρηθεί, ε, να δουλέψουμε πάνω στην αναθεωρημένη ε, οδηγία για την άδεια μητρότητας, η οποία οδηγία ερίζεται πάνω σε δύο πυλούν, πυλώνες. Να επεκταθεί η διάρκεια της άδειας από τις 18 από τις 14 στις 18, αν, όχι και 20 εβδομάδες, και αυτό είναι το ιδανικό, και επίσης ε, θα πρέπει ιδανικά η οδηγία να θεσμοθετεί τουλάχιστον δύο εβδομάδες ε, άδειας πατρότητας, με ε, βεβαίως... Ε, ε, ανταμοιβή, με να συνεχίζεται ή, πληρω, ή μη το μισθό του εργαζομένου κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου. Και μάλιστα θα έλεγα ότι ο τρόπος με τον οποίο ενσωματώθηκε η οδηγία ε, σίγουρα γύρει αφιβολίες και ίσως γι' αυτό το λόγο δεν συμμορφώθηκαν και κάποιες χώρες ή δυσκολεύτηκαν να το κάνουν. Τώρα, ως προς τα νέα εργαλεία, π.χ. τις ειδικέ συστάσεις αναχώρα βάσει του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, θα πρέπει αυτά να αξιοποιηθούν για να γίνεται σωστή παρακολούθηση και εποπτεία και τέλος, ως προς τους στόχους της Βαρκελόνης, νομίζω ότι το Συμβούλιο θα πρέπει και θα προσπαθήσει να επιβεβαιώσει τους στόχους αυτούς και να εξετάσει πιο μακροπρόθεσμους στόχους για τη φροντίδα ή σε βάθος χρόνου και όχι μόνο την φροντίδα των παιδιών σε μικρή ηλικία. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ε, Ντορότα Σέλεβα γιατί με την εισήγησή ε, μας ε, βοήθησε σε εμά τους βουλευτές που εργαζόμαστε εδώ καθημερινά να αντιληφθούμε ότι η προσπάθειά μας κυρίως για τα επόμενα χρόνια είναι να υπάρχει μια, σε νέους χαρακτήρας με τον οποίο θα αντιμετωπίζεται αυτό το θέμα και στις διάφορες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενίος χαρακτήρας λοιπόν και αυτό μπορεί να γίνει μόνο με την καθημερινή μας εργασία και θα πρέπει να είμαστε σίγουρα θα το κάνουμε η προσπάθειά μας για τα επόμενα χρόνια γιατί και στην προηγούμενη θητεία ήμουν παρούσα και δώσαμε μεγάλη μάχη για την άδεια μητρότητας και επίσης για την άδεια πατρότητας. Όπως το είπε, εσύ, είναι η κατάσταση ενός διαφορετική από τη μία χώρα στην άλλη. Πάνω χάρη ισχύει στην Ιταλία, αλλά κανείς δεν το χρησιμοποιεί με μία έρευνα ίσως ε, ένας άνδρας ε, από εδώ και από εκεί είχε αυτή την άδεια πατρότητας και κυρίως εσύ μίλησες για το πώς θα συμφιλειωθεί ο χρόνος που αφιερώνεται στην εργασία και ο χρόνος που αφιερώνεται στην οικογένεια. Πολύ σωστά το είπες ότι τα τελευταία χρόνια και με συγχωρείς που μιλάω στον ελληνικό είμαστε κοντινές στην ηλικία και αυτά τα τελευταία χρόνια βέβαια οι γυναίκες ε, απασχούνται περισσότερο στην εργασία, αλλά όχι όμως των μητέρων και εκείνες που θέλουν και πάλι να επανεφανιστούν μετά από την εγκυμοσύνη τους ε, και τη μητρότητά τους στο χώρο εργασίας. Θα πρέπει να εργαστούμε ώστε να δώσουμε τα δίκαια, τα σωστά εργαλεία στις γυναίκες και στην οικογένεια. Όταν λέμε ότι θέλουμε να υποστηρίξουμε τη γυναίκα, υποστηρίζουμε την οικογένεια ουσιαστικά. Σε ευχαριστώ λοιπόν για όσα μας είπες και κυρίως για την γενικά την εισήγησή της σου. Υπάρχει διάθεση νομίζω να υποβληθούν ερωτήσεις στην Τωρότα Σέλεβα για να δούμε. Μήπως η συνάδελφος αντιπρόεδρος θα ήθελα να λάβει το λόγο για να σχολιάσει την παρέμβαση της εισηγητριάς μας. Όχι. Καμία ερώτηση. Τίποτα. Καμία. Τι να κάνουμε. Υπέροχα. Πάμε παρακάτω. Σας ευχαριστούμε. Πάμε τώρα στο δεύτερο μέρος της συνάντησή μας. Οι γυναίκες στην πολιτική και στην οικονομική διαδικασία λήψεων αποφάσεων θα αναλάβει μία συνάδελφος την Προεδρία στο δεύτερο αυτό μέρος της συναντησής μας. Σας ευχαριστώ για μέχρι τώρα. Θα μιλήσω πορτογαλικά. Καλό απόγευμα. Είμαι αντιπρόεδρος της Επιτροπής Δικαιωμάτων της Γυναίκε και Ίσων Ευκαιριών. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι εδώ και προεδρεύω στη συνάντησή μας. Είναι πολύ σημαντικό σήμερα το θέμα αυτό εμείς κάνουμε μία εκτίμηση του τι ακριβώς γίνεται και μάλιστα με τέτοιο τρόπο ώστε να καταλάβουμε πώς θα δράσουμε καλύτερα στο μέλλον. Για το δεύτερο μέρος της συνάντησής μας, το θέμα μας αφορά τρία κύρια σημεία, τα θεμελιώδη δικαιώματα, την λήψη απόφασης και την εξέλιξη ανάπτυξη. Έχουμε προσκαλέσει λοιπόν διάφορους συζητητές τις γυναίκες στην ε, διαδικασία λήψεων αποφάσεως πολιτικά και οικονομικά Ελεονόρ Λεπινάρ καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Λοζάνης για κοινωνικά θέματα ε, στο Ινστιτούτο των φίλων ε, διάφορες έρευνες, ε, εργασίες ε, για κοινωνικές μελέτες, νομικές, φεμινιστικό κίνημα κλπ. Θα θέλαμε λοιπόν να καλωσορίσουμε την Ελεονόρ Λεπινά και έχει το λόγο. Θα ήθελα να την ευχαριστήσω. Για 10 λεπτά λοιπόν έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ. Χαίρομαι ιδιαίτερα με τιμά που με έχετε προσκαλέσει. Θα σας μιλήσω για το θέμα των γυναικών στην διαδικασία λήψης αποφάσεων. Από το τέλος της δεκαετίας περίπου του 1980, όλο και περισσότερο έχουμε συνειδητοποιήσει τη σημασία του θέματος αυτού για τη συμμετοχή των γυναικών ε, εκεί που λαμβάνονται αποφάσεις, κυρίως σε διεθνές επίπεδο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και διαθέτουμε συστάσεις και διεθνώς που υποστηρίζουν μια μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών στους χώρους αυτούς. Σήμερα όμως με λιγότερο από 22% των γυναικών στα κοινοβούλια σε παγκόσμιο επίπεδο υποεκπροσωπούνται οι γυναίκες εκεί όπου λαμβάνονται πολιτικές αποφάσεις ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι για τα κοινοβούλια 28%, κάπως καλύτερα από ότι ο διεθνής μέσος όρος, αλλά κάτω από το 1 τρίτο, το 33 γυναικών, όπως μας είχαν υποσχεθεί το 1990 και το 1995 στη συνδιάσκεψη του ΙΕ για τις γυναίκες. Να που πάνω από 20 χρόνια μετά δεν τα καταφέραμε να πετύχουμε το στόχο όπως είχε καθοριστεί. Οι ποσοστώσεις αυτές δυστυχώς αποτέλεσαν πια ένα μηχανισμό διαδομένο, αποτελεσματικό για να αποφύγουμε παρόμοιες καταστάσεις, να τις αντιμετωπίσουμε. Και εδώ ισχύει σε διάφορα επίπεδα, διαπιστώνουμε, έχουμε περίπου 100 χώρε στον κόσμο που εφαρμόζουν με τον άλλον τρόπο ποσοστό στην πολιτική 56 ακριβώ χώρε που εφαρμόζουν ε, μέσω νόμου, δηλαδή δεσμευτικά αυτή την ποσόσταση και επίση ένα κατόφλι ποσοστώσεων που αυξάνονται και ε, περίπου ήταν το 1 τρίτο, τώρα όλο και περισσότερο πηγαίνει στο 40 και στο 50% αυτή η εκπροσώπηση, αυτή η ποσόστοση και επίσης ισχύει ευρύτερα σε διάφορα όργανα και από πολιτικής πλευράς βλέπουμε όμως και από οικονομικής σε διάφορες διεθνείς οργανισμούς εθνικούς οργανισμούς έχουμε την εφαρμογή των ποσοστώσεων διάφορες ποσοστώσεις διάφορες μορφές σημαντικό είναι να θυμόμαστε επειδή βάζουμε κατά το καπέλο το ίδιο πράγμα, διαφορετικά πράγματα είναι χωρίς κυρώσεις ποσοστό, εντάξει, εθελοντικά, σε ορισμένα πολιτικά κόμματα που λένε ότι για την ιστορική τους οργάνωση, της υποψηφιότητας ισχύει αυτή η ποσόστοση και επίση για διοικητικά συμβούλια. Εκεί υπάρχει μια νομοθεσία, αλλά χωρίς και επιβολή κύρωσης, εντάξει, είναι στην ε, διάθεση αυτών και οι σκληρές ποσοστώσεις με κυρώσεις δηλαδή μέσω νόμου συχνά και εκεί υπάρχουν κυρώσεις πάνω χάρη ε, να μην ε, γίνει δεκτό ένα ψηφοδέλτιο επειδή δεν ε, σέβεται το θέμα αυτών των ποσοστώσεων είτε ένα διοικητικό συμβούλιο να μην εισέχει επειδή δεν σέβεται αυτές τις διαδικασίες αυτή την ποσόστοση. πράγματα λοιπόν στην Ευρώπη βρίσκουμε διάφορες μορφές ποσοστώσεων Πολλά κρατημέλη εφαρμόζουν αυτές τις ποσοστώσεις και σε οικονομικό επίπεδο και σε πολιτικό επίπεδο. Κάτι σημαντικό, πολλά κρατημέλη, αυτό δεν το γνωρίζουμε, που ακόμα και στο δημόσιο, το public ε, quotas ε, που ισχύουν για τον ορισμό υπαλλήλων, είτε στο είτε στην Υπουργεία, είτε ποσοστώσεις που έχουν να κάνουν με επιτροπές οι οποίες διορίζονται από το Κοινοβούλιο, από την κυβέρνηση και αυτό το συναντούμε σε αρκετές βόρειες χώρες, χώρες του Βορρά είτε και στην Αυστρία. Και επίσης διάφορες ποσοστώσεις ε, διαφορετικής μορφής ε, για άλλους φορείς που χρηματοδοτούν το δημόσιο όπως τα πανεπιστήμια και πρωτοβουλίες στη Γερμανία ώστε να ισχύουν στα διάφορα κλάδους, στην ιατρική, στην ε, δημοσιογραφία, να ισχύουν επίσης ποσοστώσεις. Τα ισχυρά σημεία αυτών των ποσοστώσεων ποια είναι, γιατί χρησιμοποιείται αυτή η μέθοδος, επειδή λειτουργεί, τα πάει καλά. Γιατί έτσι έρχονται γυναίκες, ε, μπαίνουν γυναίκες σε αυτούς φορείς από εκεί που αποκλειόταν κανονικά. Το 2012, παραδείγματα, στις 10 χώρες στον κόσμο που είχαμε την υψηλότερη αύξηση συμμετοχής στο Κοινοβούλιο Γυναικών, οι, νέα, χώρε 9 χώρες στις 10 εφάρμοζαν την ποσόστοση. 6 στι 16 χώρες ε, στην Ευρώπη που υπάρχουν περισσότερες γυναίκες εφαρμόζουν ε, μια ποσόστοση μέσω επιβολής νόμου. Και οι ποσοστώσει ε, αποτελεσματικέ είναι ιδιαίτερα σε χώρε που ιστορικά σημείωνα μια ισχνή παρουσία γυναικών όπως η Ισπανία, Γαλλία, Πορτογαλία, Βέλγιο, Πολωνία ή και Σλοβενία. Τι βλέπουμε ότι με τις ποσοστώσεις έχει μεταβληθεί γοργά η κατάσταση και ποσοτικά έχουν αυξήσει ιδιαίτερα οι γυναίκες στη Σλοβανία από το, σε 12 χώρες από 12 πήγαμε στις 34 γυναίκες στην Νορβηγία στα δικαιωτικά συμβούλια σε 6 χρόνια από το 6% γυναικών πήγαμε στο 40% γυναικών Ωραία λοιπόν είχαμε ποσοτικά άλματα ιδιαίτερα όταν ακριβώ έχουμε να κάνουμε και με κυρώσει που επιβάλλονται αν δεν γίνονται σεβαστά αυτά για τις ποσοστώσεις, για την πολιτική είτε για οικονομικού κλάδου, ακριβώ είναι αποτελεσματικέ. Βέβαια, κατά πορεσμένε συνθήκες, όπως συμβαίνει πάντα. Στην πολιτική σημαντικό είναι ιδιαίτερα γιατί παρατηρούμε ότι οι ποσοστώσεις αυτές ε, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν και στα ψηφοδέλτια για το ποια θέση καταλαμβάνουν στο ψηφοδέλτιο. Γιατί οι ποσοστώσεις που δεν λένε τη σειρά ε, τελικά οι γυναίκες μπαίνουν κάτω-κάτω στο ψηφοδέλτιο, άρα λοιπόν δεν εκλέγονται. Άρα λοιπόν μπορεί να έχουμε με 30-40% ε, συμμετοχή, αλλά δεν καθοριστεί και ποιες θέσεις θα έχουν πάνω-πάνω ή κάτω-κάτω, τότε δεν έχει καμία σημασία αυτό. Αυτό πασγαρί έγινε στην Πολωνία, συνέβη στην Πολωνία. Με κάποια άλλη συνθήκη θα πρέπει να είναι ένα κατόφλι και όχι μια οροφή υπό το ιστόστοση το 33%-25% δημιουργούν πρόβλημα αυτές οι ποσοστώσεις γιατί είναι η ενότητα ορφή και όχι κάτι που βοηθάει τον αύξηση των αριθμών των γυναικών όπως στη Γαλλία ή στο Βέλγιο πριν να προβεί σε αναθεώρηση του νόμου ε, λιμνάζουν αυτοί οι αριθμοί σε ποσοστά ιδιαίτερα χαμηλά. και όμως και κυρώσεις διαφορετικά δεν είναι αποτελεσματικές ε, ποσοστώσεις επίση, ένα έλεγχο να γίνεται για να δούμε ότι πραγματικά εφαρμόζονται αυτέ οι ποσοστώσεις. Σημαντικό είναι γιατί ε, ο έλεγχο ε, δίνει αποτελέσματα και όταν υπολογίζουμε τον αριθμό των γυναικών βλέπουμε πού ακριβώς δεν ε, προχωράει η κατάσταση, βλέπουμε για τα προβλήματα, πού παραμένουν τα προβλήματα και έτσι μπορούμε να επεξεργαστούμε μια νέα νομοθεσία για να αποφύγουμε το πρόβλημα. Να λοιπόν που δημιουργεί κάτι το θετικό σαν κύκλο. Αντίθετα, το πώς μπορεί κανείς εθελοντικά να το κάνει πάνω στα διάφορα κόμματα. Αυτό είναι προβληματικό μερικές φορές. Ορισμένα κόμματα εφαρμόζουν, πως τόσο άλλα όχι κυρίως της αριστεράς αλλά και αλλού δεν εφαρμόζονται όπως πρέπει δίκαια και η αποτελεσματικότητα είναι χαμηλότερη στην Αγγλία, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μόνο οι εργατικοί εφαρμόζουν μια ποσόστοση. Τι προκαλεί αυτό. Ε, πάνω από το 84% των γυναικών που εκλέγονται στο κοινοβούλιο είναι στο εργατικό κόμμα και είναι περίπου 24% το ποσοστό γυναικών γενικά στο Βρετανικό Κοινοβούλιο. Δεν αυξάνει εδώ και πολλά χρόνια. Και παραλαμβάνομαι, οι περισσότερες γυναίκε που εκλέγονται μπροστά είναι από την αριστερά. Για τους του οικονομικού τώρα. Αυτή ε, εθελοντικά που ενθαρρύνονται οι επιχειρήσεις να συμπεριλάβουν στο δίκαιο του Συμβούλιο γυναίκες και θέλουμε να μάθουμε τελικά το γιατί όπως στην Ισπανία και στη Δανία αλλά τα μέτρα αυτά τελικά δεν αποδίδουν απλά και μόνο εξηγήστε μας γιατί δεν συμμετέχουν δεν φτάνει λοιπόν αυτό δεν αυξάνει ο αριθμός των γυναικών που συμμετέχουν θα πρέπει να δούμε τώρα για τις ποσοστώσεις τι άλλο προκαλεί να δούμε και τα υπόλοιπα θετικά σημεία, πτυχές που είναι σημαντικές. Μία από τις σημαντικές πτυχές ε, είναι το να αποφύγουμε τις διακρίσεις απέναντι στις γυναίκες σε ορισμένα όργανα γιατί όταν έχουμε μια ποσόστοση ασχολούμαστε περισσότερο με το να ξέρουμε τι γίνεται. Έχουν τα προσόντα, θέλουν να συμμετάσχουν στην πολιτική αυτές οι γυναίκες, έχουν πραγματικά διάθεση να εργάζονται και θέλει κανείς να ξέρει ποιος είναι ο θεσμικός ε, χαρακτήρας ε, που είναι εις βάρος των γυναικών είναι και ποιος υποεκπροσωπείται μέχρι τώρα. Άρα λοιπόν ιδανικά η εφαρμογή προς εντάξει θα μπορούσε κανεί να αλλάξει την πρόσληψη όπω και την, εντονισμό να διευκρινιστούν τα πράγματα πώ προχωράει κανεί, να δούμε καλύτερα τι δεξιότητε, τα προσόντα και να αλλάξουμε ενδεχόμενα τα κριτήρια αυτά και έτσι να παρακάμψουμε εμπόδια. Και στον πολιτικό κόσμο ξέρουμε ότι με ίσες δεξιότητες προσόντα οι γυναίκες ε, δεν επιλέγονται από τις περισσότερο από τους άνδρες ε, ή όπως τους άνδρες ε, για τις θέσεις αυτές λοιπόν ενώ έχουν τα προσόντα πετυχαίνουν λιγότερα πράγματα γι' αυτό χρειάζεται ένας μηχανισμός δεσμευτικός ώστε να δούμε ποιες είναι οι γυναίκες αυτές και να μπορέσουν να υποβάλουν υποψηφιότητα Αυτά. Κάτι ακόμα θετικό για τις ποσοστώσεις. Ποιο είναι τη κατάπνιση να την πούμε έτσι, μάλλον δεν τι διαπιστώνουμε και στην πολιτική αυτό πράγμα όπου τε διοικητικά αυτά καθήκοντα, τα υπουργεία καθήκοντα πηγαίνουν σε διαφορετικό κόσμο και να δούμε υπάρχουν σημαντικά που εφαρμόζονται για τον ορισμό ας πούμε σε υπουργικές επιτροπές στις βόρειες χώρες και έτσι γίνεται δεν είναι αρκετά ομοιογενές το, το, το, το, η σύνθεση και είναι θα πρέπει να δούμε ότι μερικές φορές ε, λόγω της διάκρισης αυτής δεν υπάρχει κατάλληλη συσπήρωση. Κάτι ακόμα για να δούμε ποιος είναι ο ρόλος πρότυπο κυρίως για τις νέες γυναίκες και επίσης να προχωρήσουμε σε μια διαφοροποίηση για τα όργανα που λαμβάνουν αποφάσεις για τα δικαιωτικά συμβούλια στη Γαλλία από τη στιγμή που ισχύει αυτό τα δικαιωτικά συμβούλια ανανεώθηκαν και ακόμα περισσότεροι ε, που δεν είχαν πείρα μέχρι τώρα αλλά και που έχουν ε, προερχονται και από το εξωτερικό. Αυτό για τα διοικητικά συμβούλια. Σημαντικό όμω είναι κάτι να σημειώσουμε ότι δεν μπορούν να πετύχουν τα πάντα οι ποσοστώσει εντάξει, να σπάσουμε δεσμά, να αποφύγουμε εμπόδια κατά των διακρίσεων. Δεν μπορούν να αλλάξουν όμω τα πάντα. Έχουμε κάτι το καινούριο επίσημο που επιτρέπει βέβαια κάτι το καινούριο στις γυναίκες. Ταυτόχρονα όμως ε, δεν ε, αποφεύγουμε, δεν παρακάπτουμε και όλα αυτά που ισχύουν άτυπα σε ένα σε ένα όργανο ο οποίος αποκλείει τις γυναίκες ε, και θα επανέλθω σε αυτό, θα δει και τις συστάσεις στη σελίδα 12 της έκθεσης. Τι σημαίνει ότι θα πρέπει μαζί με τις ποσοστώσεις να συνδευτούν και από διάφορα μέτρα για να αλλάξει η αντιμετώπιση πραγματικά, η νοοτροπία και να δούμε για τη συμμετοχή των γυναικών τώρα στα όργανα λήψης αποφάσεων. Υπάρχει μια κάποια στιγμή που σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ας πούμε την πρόταση οδηγίας του κ. Ρέντινγκ το 2012, και υπήρξε αντίθεση από τη Γερμανία, μια κάποια αντίθεση, εντάξει κανονικά δεν εκφράζεται πλέον. Νομίζουμε ότι η Γερμανία μέχρι το τέλος του 2014 θα θέσει ισχύ μια ποσόστοση για το Δικαιωτικό και υπάρχει μια κάποια παρόμοια στιγμή αυτή η σημερινή που είναι υπέρ νομίζουμε της ε, υιοθέτηση σημαντικών μέτρων, δεσμευτικών μέτρων πάνω στο θέμα αυτό είναι βασικός παράγων αυτά η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω οδηγιών και συστάσεων αλλά επίσης σημαντικός παράγων γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει διάφορους τοπικούς φορείς, οργανώσεις υπέρ των ε, γυναικείων δικαιωμάτων που έχουν κινητοποιηθεί ιδιαίτερα στην οικοεπίπεδο επίπεδο για τη θέση ισχύ αυτών των ποσοστώσεων και δικτύων εμπειρογνωμών, πολύ σημαντικό σε διάφορες χώρες ώστε να υπάρξουν νόμοι που να επιτρέπουν θετικά πολιτικέ δράσει υπέρ των γυναικών, να χάρη στην πολιτική και είναι πολύ σημαντικό να συνεχιστεί από την εργασία. Το θέμα που τώρα είναι να ξέρουμε σε ποιο σημείο μια οδηγία που θέτει ισχύ σε ένα δικαιωτικό συμβούλιο μια ποσόστοση θα περνούσε ας πούμε το τεστ του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου γιατί νομίζω περίπου τα μέσα του 1995 είχαμε κάτι το θετικό παρά το ότι όλα αυτά από το 1976 είναι στις ευρωπαϊκές συνθήκες αλλά το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ε, περιορίζει τις ε, όρους εφαρμογής ε, με αποφάσεις που τελικά επιτρέπουν τις ποσοστώσεις. Δεν θα πρέπει να θεωρούμε ότι η αντίθεση είναι τόσο ισχύρη ώστε να, μπορέσει να αποφύγει την εφαρμογή ποσοστός. Για να δούμε τι μπορεί να κάνει κανείς. Να δούμε είναι τα πολιτικής πλευράς. Δεν μπορούν να πετύχουν τα πάντα. Χρειάζονται και συνδευτικά μέτρα να ενθαρρύνουμε τα πολιτικά κόμματα το κάνουμε και επίσης με εσωτερικές ποσοστώσεις εκεί και στις υποψηφιότητες τους, στα ψηφοδελτιά τους να υπολογίσει κανείς τον αριθμό των γυναικών, την παρουσία τους στα διάφορα όργανα ταυτόχρονα όμως και διαφορετικά εργαλεία ιδιαίτερα σημαντικά. Τα μέτρα αυτά που δεν είναι ποσοστώσεις θα μπορούσαν να ισχύσουν και εθελοντικά από τα κόμματα. Ταυτόχρονα όμως και να επιβληθούν. Να επιβληθούν μέσω κατάλληλης ρύθμισης, ε, ε, ρύθμισης και επιβολής με δημόσιο χαρακτήρα. Θα πρέπει να δούμε το πώς ε, στο καταστατικό θα μπορούσε να ενό να αναγνωριστεί η ισότητα ανδρογυναικών ότι πρόκειται για σημαντική κύρια αξία και επίσης ε, ότι μπορεί κανείς να ρυθμίζει, πρέπει να ρυθμιστεί στις ε, εκλογές, στις προεκλογές η παρουσία γυναικών και στα μέσα και μια ενημέρωση για τις γυναίκες στα πολιτικά κόμματα, όχι μόνο μόνο για τις γυναίκες και μια εκπαίδευση για τα δύο φύλλα και να αποφύγει κανείς τις διακρίσεις λόγω φύλου. Επίσης κάτι θα μπορούσε να επέμβει στο ε, εσωτερικό κανονισμό χρηματοδότησης ε, σχετικά με τον ορισμό ή πώς θα οριστεί κάποιος υποψήφιος. Επίσης ε, στα κόμματα όπως και υπάρχει σύσταση θα μπορούμε να το κάνουμε αυτό από τα μέσω των εθνών να προωθήσουμε τα γυναικεία δίκτυα στα πολιτικά κόμματα. Αυτά για τα εθνικά κοινοβούλια όπως το είπα, μπορεί κανείς να ρυθμίσει νομοθετικά όλα αυτά που μόλις είπαμε και για τη χρηματοδότηση τη δημόσια στα πολιτικά κόμματα σχετικά με αυτά που υιοθετούν και τα Εθνικά Κοινοβούλια θα πρέπει να υιοθετούν ε, διάφορες ποσοστώσεις και για την πολιτική και για την οικονομική επιτυχία στο δημόσιο και επίσης την κάλυψη των μέσων ενημέρωσης των προεκλογικών στρατιών. Είναι σημαντικό και αυτό μπορεί να γίνει μόνο σε επίπεδο εθνικών κοινοβουλίων να ε, επαναξετάσει το μηχανισμό για τις συνταξιδοτήσεις πανσχαρή βουλευτών ε, όλων των εκπλεγμένων ε, γιατί μια εναλλαγή γυναικών ε, αυτό ισχύει για τις γυναίκες κυρίως ε, για βραχύτερα χρονικά διαστήματα κλαίγονται από ότι άνδρες ε, και πολλές φορές σε εισαγωγικά αποβάλλονται και τι θα κάνουν, πώς θα επανέλθουν στην εργασία τους τη θητεία τους, πώς επηρέασε την εργασία τους, όλα αυτά τα πράγματα. Όλα αυτά ίσως τους αποτρέπει από το να είναι υποψήφιες και να ακολουθήσουν μια πολιτική καριέρα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό να μπορέσει κανεί να βελτιώσει τον όλο, το όλο θέμα πάνω χάρη των συντάξεων για τους βουλευτές και πώς μπορούν να επανέλθουν στην αγορά εργασίας ε, και στο τέλος πώς γίνεται ένα απολογισμό των δεξιοτήτων και από τα μέτρα που μπορούν να εφευθούν από τα Εθνικά Κοινοβούλια έχουμε και το ότι μπορεί κανείς να συμπληρώσει πολύ σημαντικό τις ποσοστώσεις αυτές πάνω χάρη για τα διοικητικά συμβούλια και αυτό να υπάρχει μια υποχρέωση να συντάσσεται μια αιτήσια έκθεση που έχει να κάνει με τις ευκαιρίε σε μια εταιρεία, μια επιχείρηση και ένα σχέδιο ε, πενταετές ε, για τα επόμενα πέντε χρόνια με τα δύο φύλλα για την ισότητά τους. Αυτό που κάνουν και οι Γάλλοι ψηφίστηκε αυτό το 2011 για τα δικαιωτικά συμβούλια και υπάρχει μια υποχρέωση ετησίως να ψηφίζεται από το, συμβούλιο, από το Διοικητικό Συμβούλιο μία έκθεση σχετικά με την ισότητα σε αυτή την εταιρεία για όλες τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν παρόμοια υποχρέωση σύμφωνα με τον νόμο να έχουν μια ποσόστοση στο Κεντρικό Συμβούλιο. Έτσι να κάνει μια εκτίμηση των ποσοστώσεων σε, στα υψηλότερα σκαλιά με τις ευκαιρίες παντού και έτσι να μπορέσει να μπορέσουν να ωφεληθούν όλοι από τις ποστώσεις αυτές ε, για τους ε, εργαζόμενους. Πρόκειται λοιπόν για μια μεταρρύθμιση ιδιαίτερα σημαντική. Και όπως άλλωστε είπε η προηγούμενη ομιλήτρια, Σημαντικό είναι να συμπληρωθούν όλες αυτές οι μεταρρυθμίσεις αλλαγές με κατάλληλα μέτρα που να είναι υπέρ κυρίως της αδιασπατρότητος, ε, θα πρέπει να είναι να μπορέσουν και οι γυναίκες ε, να ασχοληθούν με τις αποφάσεις ακριβώς και οι άνδρες να συμμετέχουν στον τομέα αυτό. Και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τελειώνοντας, ε, παίζει ένα σημαντικό ρόλο για να μπορέσει κανείς ε, να συνεχίσει να βοηθάει, να υπάρξει μια συνειδητοποίηση, επειδή υπάρχει αυτό το θέμα της εκπροσώπησης γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων και να το κάνει αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέσω καταλήνων εκθέσεων να ενθαρρύνει αυτή την αναγνώριση των θετικών δράσεων ενεργειών ε, από το 76 ήδη στις συνθήκες υπάρχουν, αλλά δεν τις αναλαμβάνεται κανείς όπως πρέπει ότι είναι κάτι το συμπληρωματικό. Ε, νομίζουν ότι είναι κατά της ε, ε, αντιμετώπισης. Θα πρέπει να καταλάβει κανείς ότι η ποσοστός μας χάρη είναι κάτι το συμπληρωματικό στα νόμιμα μέσα τα οποία υπάρχουν και ισχύουν για να ισχύσει πράγμαση αυτή η ισότητα και να υποστηρίξει κανείς σίγουρα και την πρόταση της Επιτροπής για ποσοστώσεις στα διοικητικά συμβούλια στην Ευρώπη, αλλά να προσέξουμε κάτι. Να εφαρμόζεται αυτές οι ποσοστώσεις όχι μόνο στα μέλη που έχουν εκτελεστική εξουσία, αλλά και, εκείνους, αλλά και σε εκείνους που δεν έχουν. Στη Γερμανία, τι παρατηρούμε. Εάν εφαρμοστεί σε εκείνου που δεν έχουν μια εκτελεστική εξουσία, τότε θα έχουμε γυναίκες μόνο εκεί και όχι εκεί που πραγματικά λαμβάνονται αποφάσει στα διοικητικά συμβούλια. Σημαντικό είναι λοιπόν οι ποσοστό αυτέ να εφαρμόζονται παντού για όλα τα διοικητικά συμβούλια πάση φύσεως και να υπάρχει μια πραγματική ισότητα με μια κατάλληλη έκθεση ετήσια το πώ εφαρμόζονται όλα αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα μπορούμε να κάνουμε μια σύντομη συζήτηση. Οι ευρωβουλευτές που είναι στην αίθουσα, παρακαλώ, έχετε κάποια σχόλια να κάνετε ή κάποια ερώτηση που θέλετε να θέσετε. não havendo nenhuma questão, eu vou colocar uma questão. Από ό,τι βλέπω δεν υπάρχουν ε, ερωτήσεις, όμως θα ήθελα και εγώ από την πλευρά μου να πω ε, κάτι. Θα μιλήσω αργά ε, για τους διερμηνείς, λέει η ομιλήτρια. Όταν γίνονται μελέτες για τα συστήματα ποσοστώσεων, και δεν έχω διαβάσει τη μελέτη για την οποία μιλάτε, υπάρχουν ιδέες σχετικά με τον χαρακτηρισμό των κοινωνικών τάξεων από τις οποίες προέρχονται οι άνθρωποι που επηρεάζονται από το σύστημα των ποσοστώσεων. Φυσικά φαίνεται ότι πρέπει να γίνει μια ευρύτερη συζήτηση όχι μόνο για τις διακρίσεις κατά των γυναικών, αλλά και για τις διακρίσεις σε σχέση με την οικονομική θέση των γυναικών. Θα ήθελα να ακούσω κάτι γι' αυτό, αν γίνεται. Ναι, σας ευχαριστώ. Υπέροχη ερώτηση. Όταν μιλάει κανείς για τους χώρους που λαμβάνονται οι αποφάσεις ε, κυρίως ε, από την κοινωνική ελίτ ε, άνδρες γυναίκες τι διαπιστώνουμε για το γαλλικό νόμο για τις προστώσεις στα διοικητικά συμβούλια. Τι παρατηρούμε. Οι γυναίκες έχουν τα ίδια κοινωνικά και επαγγελματικά χαρακτηριστικά όπως και οι άνδρες που συμμετέχουν εκεί. Είναι μια μικρή ελίτ ε, ηγετική ομάδα. Οι ποσοστώσεις κάπως αλλάζουν τα χαρακτηριστικά αυτά, τα κοινωνικά και επαγγελματικά χαρακτηριστικά. Ας πούμε τους βουλευτές. Υπάρχει ένα προφίλ κάπως διαφορετικό, μια εικόνα διαφορετική, με γυναίκες που θέλουν να συμμετάσχουν στην πολιτική και που προέρχονται από το δημόσιο και που εργάζονται σαν ε, δασκάλες ή καθηγήτριες, καμιά φορά είναι και κοινικοκύρες. Κάτι που δεν το παρατηρούμε στις άνδρες ε, που είναι γιατροί, δικηγόροι, παρόμοια επαγγέλματα οι άνδρες. Λοιπόν, αυτά τα... Υπάρχει μια κάποια μικροδιαφοροποίηση χάρη την ε, συμμετοχή των γυναικών. Αλλά η εικόνα των εκλεγμένων ε, δεν είναι αντιπροσωπευτικό όπως, ο υπόλοιπος πληθυσμό. Το ίδιο εικόνα γυναικών επίσης ε, έχει κάτι βοηθιέται. Θα πρέπει να δούμε αυτά τα μέτρα πώς θα συνδεθούν με ενεργά μέτρα υπέρ της ισότητας στο σύνολο, στο middle management, στους εργαζόμενους, ώστε να εφαρμοστεί και οι άλλες γυναίκες και όχι μόνο εκείνες που είναι σε αυτή την ε, ηγετική κατηγορία, την πάνω-πάνω. Ευχαριστώ. Από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Πώς... Στο επόμενο θέμα μας, στην επόμενη παρουσίαση, Ζήτω συγγνώμη. Υπάρχει μια ερώτηση. Ήθελα να ρωτήσω αν ανάμεσα στις συστάσεις Συνήθως, ε, ιδιωτικά όταν μιλάμε σε τέτοιες συζητήσεις λέμε ότι ε, δεν υπάρχουν γυναίκες επειδή δεν βρίσκουμε γυναίκες. Αναρωτιέμαι αν θα ήταν καλό να έχουμε ε, και κάποιες συστάσεις για τη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων. Σίγουρα υπάρχουν κάποιες, όμως να ενθαρρύνουμε ίσως ιδιαίτερα ε, αυτούς που ψάχνουν ταλέντα ε, για να υπάρχει πραγματικά μια στρατηγική ισότητας ε, των ατόμων ήδη από τη στιγμή του διορισμού το, επιλογής των ανθρώπων που θα μπουν σε αυτές τις θέσεις της εταιρείας. Κοιτάξτε, ε, το επιχείρημα που χρησιμοποιείται συνήθως είναι ότι όταν υπάρχουν ποσοστώσεις βρίσκονται τελικά γυναίκες. Και αυτό που διαπιστώνουμε, αν δούμε και το παράδειγμα και του γαλλικού αλλά και του νορβηγικού νόμου, ας πούμε στο γαλλικό νόμο για τα διοικητικά συμβούλια, βρήκαμε γυναίκες με ακριβώς τα ίδια προσόντα, την ίδια εμπειρία, το ίδιο υπόβαθρο. Δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα και οι εταιρείε όταν είδαν ότι μπορούν να βρουν τέτοιες γυναίκες σταμάτησαν να παραπονούνται για τον νόμο. Και αυτές με τη μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση, μεγαλύτερες δηλαδή εταιρείε είναι ήδη πέραν του ποσόστοσης για το 2014, άρα δεν είχαν κανένα πρόβλημα να βρουν γυναίκα. Από την άλλη, βέβαια, ε, έλεγαν ότι ίσως θα είναι οι ίδιες γυναίκες σε όλα τα δημοκρατικά συμβούλια. Ούτε αυτό τελικά συνέβη. Υπάρχει μια μεγάλη ποικίλια, μεγάλος αριθμός γυναικών. Άρα το επιχείρημα τελικά δεν ισχύει. Και αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι ότι όντω μπορούμε να ενθαρρύνουμε αυτούς που ψάχνουν ταλέντα, όμως αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι οι γυναίκες οι ίδιες ε, οργανώνονται και υπάρχουν αυτές οι γυναίκες οι οποίες βρίσκονται σε διοικητικές θέσεις και φτιάχνουν ένα δίκτυο με γυναίκες σε αντίστοιχες θέσεις για να υπάρχει μια δεξαμενή με ικανές γυναίκες που ε, τελικά βλέπουμε ότι με βάση τις, ποσοστά, τις ποσοστώσεις ενθαρρύνεται η ύπαρξη μιας σειράς δικτύων. Υπάρχει μια ευαισθητοποίηση και βρίσκουμε γυναίκες για αυτές τις θέσεις. Ικανές. Ε, ε, eh, Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις από την αίθουσα, από κάποιον που έχει κάποιο σχόλιο ή ερώτηση. Εσείς εκεί πίσω, παρακαλώ. Can you hear me? Με ακούτε? Δεδομένης αυτής της ιδέας των ποσοστώσεων, εγώ είμαι ε, διπλής εθνικότητας ε, και Βέλγιο, άρα το θέμα των ποσοστώσεων είναι ένα καυτό θέμα συνήθως. Ένα θέμα ε, δύσκολο και για μένα την ίδια, γιατί αναρωτιέμαι πώς ε, κανείς θα ασχολείται με το θέμα των ποσοστώσεων για γυναίκες που ε, είναι ε, ας πούμε ε, από και γενικά αν υπάρχει και κάποια πολιτιστική ας πούμε διάκριση σε σημείο που ακόμα και οι έγχρωμοι ε, μπορεί τελικά να βρίσκονται σε μενεκτική θέση γιατί θα υπάρχει κάποιο πέναλτι, κάποια τιμωρία για αυτού. Θα μπορούσατε να πείτε κάτι για αυτό το θέμα. Ναι, σημαντικό είναι. Δεν διαθέτουμε ιδιαίτερε μελέτε για το πώ επιδρούν οι ποσοστώσει στι εθνικέ μειονότητα, αλλά υπάρχουν λίγε και θα το δείτε, αναφέρονται στην έκθεση μα, άρα για το Βέλγιο. Τι παρατηρούμε. Σχετικά με θέματα πολιτική, οι ποσοστώσει είναι υπέρ των γυναικών που πρόκειται από εθνικές μειονότητες και το ίδιο πιστώνεται και στη Γαλλία τουλάχιστον ε, σε επίπεδο τοπικών εκλογών, δημοτικών εκλογών κλπ. Κοινικός υπολογισμός που λένε εντάξει μια, αφού θα βάλουμε, θα βάλουμε μια γυναίκα ας βάλουμε και μια εγχρωμή και το βλέπουμε και στις κυβερνήσεις αλλά ποσοστώσεις δεν είναι εις βάρος των γυναικών που προέρχονται από εθνικές μειονότητες ε, έγχρωμες κλπ. Δεν είναι αντίον όχι, το αντίθετο. Τώρα, το ερώτημά σας, όπως και της Αντιπροέδρου, σε αυτό στοχεύει ότι υπάρχει μια κάποια διαφοροποίηση στην ομάδα των γυναικών. Δεν αντιμετωπίζουν το θέμα όλες με τον ίδιο τρόπο. Τελικά ποσοστό θα είναι υπέρ όλων των γυναικών με τον ίδιο τρόπο. Ποια είναι η απάντηση. Όχι. Όχι. Γιατί πάνω σχετικά που λαμβάνονται αποφάσεις Καταρχά, ε, εκεί καταλαμβάνονται αυτές τι θέσεις από προέρχονται από τις ανώτερες κοινωνικές ομάδες. Ε, αλλά επαναλαμβάνω, η ποσοστό είναι υπέρ των ασθενεστέρων ε, τάξεων, αλλά τουλάχιστον ανοίγουν δυνατότητε, δημιουργούν δυνατότητε και για αρκετέ άλλε γυναίκε να συμμετάσχουν. Και αυτό για τι ποσοστώσει δεν μπορούμε να πούμε σίγουρα ότι ανοίγουν το δημοκρατικό δρόμο. Πάντως βοηθούν τις γυναίκες που προέρχονται από μειωτικές ομάδες Δεν ξέρω αν θα γίνεται καλύτερη επιλογή με κόσμο που προέρχεται από αυτές τις ομάδες για να υπάρξει ένας εκδημοκρατισμός ε, σε τόπους όπου λαμβάνονται αποφάσεις, απαιτούνται μηχανισμοί και απαιτείται μια αναδιοργάνωση διαρθωτική, μπορούμε να την πούμε, πολύ ευρύτερη. Τα διοικητικά συμβούλια, οποιοδήποτε μπορεί να συμμετάσχει εκεί, δεν νομίζω να το πετύχουμε. Αλλά για τα δικά της συμβούλια πάντως φαίνεται καθαρά το ότι υπάρχει μια συζήτηση για τις ποσοστώσεις παρόμοιες για αρκετές επιχειρήσεις ε, δεν έχει να κάνει μόνο με τα φύλλα, αλλά με τη διαφοροποίηση. Ανοίγει μια πόρτα για να πει κανεί πού να προβούμε σε μια διαφοροποίηση ανάλογα με το εθνικά προέρχοντα και όχι μόνο για τα φύλλα για τη σύνθεση του Συμβουλίου αυτού. Πάντως αυτή η συζήτηση μπορεί να ξεκινήσει για άλλα πράγματα και για άλλες μειωτικές ομάδες ε, που να συμμετάσχουν στα όργανα λήψης αποφάσεων. Ε, ελπίζω να απάντησα στις ερωτήσεις σας. Sorry, I just need follow up on that because... Συγγνώμη, θα ήθελα και να ρωτήσω για κάτι άλλο, γιατί για μια χώρα όπως η Γαλλία, όπου δεν υπάρχουν νούμερα και τεκμηρίωση για τους έγχρωμους, είναι δύσκολο κανείς να πει ότι αυτό δεν επηρεάζει ή δεν έχει αρνητικές επιπτώσεις. Ναι, Νομίζω ότι η Γαλλία είναι μια εξαίρεση που δεν πρέπει να την έχουμε ως πρότυπο. Είναι δύσκολο να κάνει κανείς γενικεύσεις βάσει της Γαλλίας. Όμως υπάρχει μια μελέτη με βάση το Βέλγιο όπου γίνονται καλύτερες μετρήσεις. Αλλά ακόμα και στην Γαλλία που δεν μπορούμε να υπολογίσουμε, μπορούμε να διαπιστώσουμε, να παρατηρήσουμε. Και στις συζητήσεις σε επίπεδο επιχειρήσεων βλέπουμε ότι όλες οι συζητήσεις που έχουν να κάνουν με το θέμα των ποσοστώσεων σε επίπεδο διοικητικών συμβουλίων για παράδειγμα αλλά και στην πολιτική στην ουσία έτρεψαν αυτή τη συζήτηση γενικότερου περιεχομένου για αυτό το κοινωνικό ζήτημα. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Ας περάσουμε τώρα στο επόμενο θέμα, το επόμενο πάνελ. Το θέμα του οποίου είναι κάτι που το Κοινοβούλιο και τα μέλη της Επιτροπής Γυναικών ε, έχουν αντιμετωπίσει ε, πολλές φορές, ε, έχουν γίνει πολλές πολιτικές συζητήσεις, έχουμε μεγάλη νομοθετική δράση σε αυτό το θέμα. Μιλάμε για την αξιοπρέπεια, την αγκαιρεότητα και την ε, πάταξη της βίας κατά των γυναικών. Έχουμε να μιλήσει εδώ μαζί μας τον Λεβαν Αλτάν, ο οποίος έχει εμπειρία στην εφαρμογή της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι νομικός σύμβουλος και σε εθνικές κυβερνήσεις αλλά και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα του δώσουμε λοιπόν... Θα του ζητήσουμε να μας δώσει κάποιες απόψεις για αυτό το θέμα. Του δίνω λοιπόν το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να μιλήσω για αυτό το πολύ σημαντικό θέμα, την αξιοπρέπεια, την ακεραιότητα και την κατάργηση της βίας κατά των γυναικών. Είναι το σημείο 4 της στρατηγικής, ήδη καλύπτεται από τη στρατηγική και έχει υπάρξει κάποια αναθεώρηση για το πώς εφαρμόζουν αυτό το θέμα ε, τα κράτη-μέλη. Επειδή έχουμε σύντομο χρόνο στη διάθεσή μας, να πω ότι θα εξετάσω λίγο το θέμα της βίας κατά των γυναικών. Θα δούμε τις ρίζες της βίας, τις ε, έμφυλες ρίζες της βίας και τον τρόπο που θα προχωρήσουμε στο μέλλον. Ε, βλέπουμε λοιπόν μια εκτεταμένη ε, φύση της βίας. Τα δεδομένα δεν είναι συνεπή, είναι λίγα, δεν γίνεται η συλλογή τους με τακτικό τρόπο. Στην Γαλλία βέβαια ε, υπάρχει πρόσφατα μια δουλειά ε, η οποία δείχνει κάποια νούμερα τα οποία μας σοκάρουν. Εκατομμύρια γυναίκες κάθε χρόνο υποβάλλονται σε σωματική και ψυχολογική βία και χιλιάδες χάνουν τη ζωή τους σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση κάθε χρόνο. Το 1 τρίτο των γυναικών σχεδόν που έχουν υποστεί, έχουν υποστεί σωματική ή σεξουαλική βία κάποια στιγμή στην ζωή τους. Αν ε, αυτό γίνει ε, ακόμη και για μια μικρή χρονική περίοδο, στην ουσία μιλάμε για 30 εκατομμύρια γυναίκες, δηλαδή ε, πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού. Τα νούμερα συνεχίζουν, αλλά αν θέλουμε να δούμε τι γίνεται με την ανθρωποκτονία, το φόνο, το 55% των γυναικών στην Ευρώπη, πέρα δηλαδή ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σκοτώνονται από τον σύντροφό τους, από την οικογένειά τους πολλές φορές. Αυτό σοκάρει και το λέμε πολλές φορές. Τι εκπροσωπούν αυτές, αυτά τα νούμερα. Μιλάμε για σεξουαλική παρενόχληση, ε, εξαναγκαστική υπάρχει ε, ε, εξαναγκασμό σε γάμο και πολλές φορές φόνο και όλα αυτά έχουν ε, ένα, μια πτυχή που έχει να κάνει με το φύλλο. Και δεν είναι απλώς βία εγκλήματα, είναι κατ' επανάληψη εγκλήματα τα οποία ε, στην ουσία πάνουν χώρα σε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Είναι πολλές φορές το αποτέλεσμα αυτής της βίας είτε σωματική σωματικά ψυχολογικά προβλήματα. Τα ψυχολογικά προβλήματα επηρεάζουν όλες τις ε, επιλογές που έχει μια γυναίκα σε επίπεδο δουλειάς, εκπαίδευσης και προοπτικών στο χώρο εργασίας. Έτσι λοιπόν όλα αυτά επηρεάζουν πάρα πολύ τη ζωή των ανθρώπων, όχι μόνο των γυναικών που είναι τα θύματα αυτών των εγκλημάτων, αλλά και των μελών της οικογένειας, των τοπικών κοινοτήτων, της κοινωνίας γενικότερα και της οικονομικής επιτυχίας της κοινωνίας γενικότερα. Πρόκειται λοιπόν για ένα πολύ σημαντικό και μεγάλο ζήτημα και αυτό έχει αναγνωριστεί. Έχει αναγνωριστεί σε διεθνές επίπεδο, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικό επίπεδο. Και έχουν ε, γίνει πολλές δεσμεύσεις από το 1979 που τα Ηνωμένα Έθνη έφτιαξαν αυτή την σύμβαση για την πάταξη των διακρίσεων κατά των γυναικών. Από τότε υπήρξαν επανειλημμένες ε, δεσμεύσεις όπως το πλαίσιο του Πεκίνου πλαίσιο δράσης ε, που επικεντρώνεται στην ε, βία κατά των γυναικών και την αντίδρασή μας σε αυτή. Επίσης έχουμε το Συμβουλίο της Ευρώπης που έχει παρέμβει για το ίδιο θέμα με την αντίστοιχη σύμβαση. Έχουμε πολλές δράσεις επίσης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό συγκεκριμένα δεν επικεντρώνεται απαραίτητα σε γυναίκες γενικότερα, αλλά μιλάμε για το εμπόριο ε, ανθρωπίνων όντων, για τη σεξουαλική εκμετάλλευση των παιδιών. Έχουμε νομοθεσία για την υποστήριξη των θυμάτων και την προστασία τους. Ε, έχουμε μέτρα προστασίας που έχουν νομοθετηθεί και το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο έχει ταχθεί υπέρ του να αντιμετωπίσουμε κάποιες από τις ε, βασικές αιτίες, από τις ρίζες αυτού του προβλήματος, έτσι ώστε να βελτιώσουμε τις ευκαιρίες για εκπαίδευση, εκπασχόληση κτλ. Υπάρχει λοιπόν δράση, πολλή δράση, πολλές δεσμεύσεις. Οι δράσεις και οι δεσμεύσεις ως τώρα έχουν επικεντρωθεί τουλάχιστον από την πλατφόρμα του Πεκίνου, του Πεκίνου ναι, και την σύμβαση της ε, Κωνσταντινούπολης έχουν επικεντρωθεί ε, σε μέτρα τα οποία είναι ολοκληρωμένα και πρέπει να είναι και συντονισμένα. Υπάρχουν τρεις βασικοί τρόποι που θα προχωρήσει κανείς. Πρώτον, η πρόληψη. Η πρόληψη του εγκλήματος. Δεύτερον, προστασία και υποστήριξη του θύματος, όχι μόνο από τη βία, αλλά προστασία και σε όλη τη διάρκεια της, των διοικητικών και άλλων ποινικών διαδικασιών, προστασία από την περαιτέρω θυματοποίηση ε, και ε, δίωξη αυτών που έχουν διαπράξει τα εγκλήματα, γιατί σε κάποια κράτη δεν είναι καν εγκλήματα ακόμα. Υπάρχουν επίσης ε, άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ανάγκη αλλαγής των πολιτιστικών ε, προοπτικών, πώς αντιλαμβάνεται κανείς τη βία κατά των γυναικών. Πρέπει να επικεντρωθούμε επίσης στην κατάρτιση και εκπαίδευση των επαγγελματιών, έτσι ώστε να συνειδητοποιήσουν ότι όντως υπάρχει βία κατά των γυναικών, να δούνε πώς θα την εντοπίζουν και πώς θα την αντιμετωπίζουν. Και τέλος έχουμε το συντονισμό, όχι συντονισμό μόνο σε επίπεδο πολιτικών, μεταξύ των πολιτικών, αλλά και στο πεδίο, γιατί η βία κατά των γυναικών επηρεάζει πάρα πολλές πτυχές της κοινωνίας. Τους οργανισμούς. Οι οργανισμοί λοιπόν που αντιμετωπίζουν αυτά τα ζητήματα θα πρέπει να είναι συντονισμένοι μεταξύ τους για να βρεθούν αποδοτικές λύσεις. Επίσης, εξετάζονται οι υπηρεσίες υποστήριξης. Πώς διασφαλίζουμε ότι παρέχεται αποτελεσματική υποστήριξη στις γυναίκες θύματα και πώς διασφαλίζουμε ότι υπάρχει ε, επανένταξη και ε, ανάρρωση από αυτά τα προβλήματα. Επίσης υπάρχουν διάφορες δεσμεύσεις σχετικά με την αποτελεσματική εφαρμογή. Υπάρχει το θέμα της χρηματοδότησης, της συλλογής δεδομένων και της παρακολούθησης. Ήδη ανέφερα την έλλειψη δεδομένων ε, που προέρχεται κυρίως ε, σχετικά από τα δεδομένα που έχουν τα κράτη-μέλη ε, σχετικά με δικαστικές παρεμβάσεις που μπορεί να γίνονται. Τέλος, έχουμε όχι μόνο έλλειψη δεδομένων, αλλά και έλλειψη παρακολούθησης, εκ των υστέρων παρακολούθησης. Από πολλές απόψεις λοιπόν βλέπουμε ότι πολλά γίνονται τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ίδιο το Συμβούλιο, έχουν ε, δεσμευθεί και έχουν ε, εκδώσει πολλά συμπεράσματα. Υπάρχουν πολλές δεσμεύσεις, αλλά όταν κοιτάμε παρόλα αυτά τις στατιστικές που υπάρχουν, βλέπουμε ότι είτε η βία κατά των γυναικών παραμένει ίδια, δεν έχει μειωθεί, ή σε κάποιες περιπτώσεις αυξάνεται. Και όχι μόνο αυτό, οι δράσεις που γίνονται είναι πολύ αποσπασματικές και είναι τελείως διαφορετικές από χώρα σε χώρα. Το ερώτημα λοιπόν είναι γιατί συμβαίνει αυτό, ποιες είναι οι διαδικασίες και οι δυσκολίες, συγγνώμη, να αντιμετωπίσουμε ένα τόσο σημαντικό ζήτημα. Για μένα είναι μάλλον το γεγονός ότι η βία κατά των γυναικών έχει μεν μια έμφυλη διάσταση, έχει να κάνει με διαρθρωτικές ανισότητες, με κοινωνικές δομές ε, του ανδρισμού. Ε, έχουν να κάνουν με το ρόλο των γυναικών και των ανδρών στην κοινωνία και έχει και επιπτώσεις στον τρόπο με τον οποίο η κοινωνία βλέπει τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίζονται οι γυναίκες και πώς οι ίδιες θα πρέπει να αντιδρούν στη βία. Αυτό σημαίνει ότι οι διαρθρωτικές ανισότητες αυξάνουν την πιθανότητα διάπραξης βίων εγκλημάτων από την πλευρά των ανδρών. Επίσης μειώνεται η πιθανότητα να παταχθεί αυτή η βία, να αντιμετωπιστεί, να αντιδράσουν τα άτομα, οι κοινωνίες, οι κοινότητες, οι τοπικές και οι κοινωνίες επίσης μειώνει τις δυνατότητες για τις γυναίκες να ξεφύγουν από αυτή τη βία, να αντιδράσουν, να μιλήσουν. Αν δείτε τις στατιστικές από την ε, έρευνα, η οποία είναι μία έρευνα πληθυσμού, δηλαδή οι γυναίκες λένε τι θεωρούν ότι συνέβη, τι πιστεύουν ότι συνέβη, δεν είναι κάποια επίσημη στατιστική από, ποινικές, από ε, θα δείτε ότι υπάρχει μεγάλη υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Τι γίνεται ε, όταν μια γυναίκα θέλει να μιλήσει, ε, πώς αντιδρούν οι ειδικοί στα προβλήματα και πώς οι άντρες θεωρούν ότι η βία είναι λύση στα προβλήματά τους. Αυτό λοιπόν που καταλαβαίνουμε είναι ότι η αντίδρασή μας πρέπει να είναι ολοκληρωμένη και συντονισμένη και μακροπρόθεσμη. Όταν ε, λοιπόν εξετάζει κανείς αυτό και βλέπει και τις διάφορες μορφές αντίδρασης που έχουν υπάρξει ως τώρα, αν δείτε τις μορφές των δράσεων που μπορεί να μας βοηθήσουν να επιτύχουμε την θετική αλλαγή, σύντο χρόνο, και τα μέτρα που μπορεί να λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση, στην ουσία μιλάμε για ε, στοχευμένες, ε, ολοκληρωμένες και συντονισμένες δράσεις για βραχυπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες δράσεις που έχουν μια συνέπεια, συμβαίνουν κάθε χρόνο για πολλά χρόνια. Δράσεις που εφαρμόζονται και παρακολουθούνται, δράσεις οι οποίες ε, ανανεώνονται, γίνονται επίκαιρες το να έχει κάνει μια ολοκληρωμένη λοιπόν προσέγγιση, να μην επικεντρώνεται μόνο σε μια μορφή βία, αλλά να εξετάζει όλες τι μορφές βία, είναι σημαντικό. Γιατί τη μία χρονιά μπορεί να μιλάμε για το εμπόριο των ανθρωπίνων όντων και την άλλη στην, ε, να επικεντρωνόμαστε στον ακροτηριασμό των γεννητικών οργάνων, αλλά αυτό δεν είναι σωστό. Πρέπει να έχουμε ολοκληρωμένη προσέγγιση, να εξετάζουμε όλα τα εγκλήματα ταυτόχρονα. Όχι να αφήνουμε το ένα τη μία χρονιά και να ασχολούμαστε με ένα άλλο. Χρειαζόμαστε όμως όχι μόνο ολοκληρωμένη δράση, αλλά και στοχευμένη δράση. πρέπει οι γυναίκες ε, να έχουν αρρωγή και βοήθεια από τις δράσεις πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα πρέπει να εξετάζουμε και την κατάσταση των διαφόρων ομάδων γυναικών, όπως αυτές από εθνοτικές μειονότητες, ε, ε, γυναίκες ας πούμε με αναπηρίες, γυναίκες με ειδικά χαρακτηριστικά, ειδικές ανάγκες και ειδικά προβλήματα που πρέπει να επιληθούν. Όλα αυτά πρέπει να τα κάνουμε ολοκληρωμένα και ε, σε όλους τους τομείς, εκπαίδευση, απασχόληση, στο δικαστικό σύστημα πρέπει να αναφερθούμε. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι χρειαζόμαστε μια ολοκληρωμένη στρατηγική για όλα αυτά. Και έχει γίνει μια τέτοια δέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν έχει πραγματοποιηθεί. Οι στρατηγικές είναι πάντοτε το καλύτερο, όμως σε κάποιες περιπτώσεις οι στρατηγικές στην ουσία δεν επιτρέπουν την, ε, τον συντονισμό. Όταν έχεις πάρα πολλές μονάδες μέσα σε μια διεύθυνση και πολλές διευθύνσεις μέσα σε ένα θεσμικό όργανο, ε, είναι πολύ δύσκολο να υπάρχει συντονισμός και να είναι συνέργειες μεταξύ αυτών. Ας πάω τώρα γρήγορα στην εφαρμογή και την παρακολούθηση. Δεν θα σας πω όλες τις συστάσεις, Έχουμε ήδη δεσμεύσει από πολλά κράτη-μέλη που έχουν υπογράψει ας πούμε, την Σύμβαση Ιστάμπουλ. Όμως ε, πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι όχι μόνο θα δεσμευθούν όλα τα κράτη-μέλη, αλλά ε, και ότι θα επικεντρώνονται στις δεσμεύσεις και θα έχουν ε, επιτυχία, θα τις επιτυγχάνουν. Και για να γίνει αυτό χρειάζονται στόχοι. Έχουμε καταφέρει σε ευρωπαϊκό επίπεδο να θεσπίσουμε στόχους για δύσκολα ζητήματα όπως η ανέχεια, η ανεργία, η πρόορη ε, παρέτηση από το σχολείο. Και δύσκολο, και βλέπουμε ότι είναι δύσκολο να γίνει κάτι τέτοιο ε, για τις γυναίκες και τη βία κατά των γυναικών. Δεν είναι εύκολο κανείς να επιτυγχάνει στόχους αλλά είναι χειρότερο να μην έχεις στόχους και να μην βλέπεις ε, εάν τελικά επιτυγχάνεις κάτι ή όχι. Βέβαια, με αυτό συνδέεται και το γεγονός ότι δεν υπάρχουν δεδομένα ούτε και δείκτες. Όλα αυτά μας περιορίζουν στη δυνατότητα παρακολούθησης. Έτσι, σε επίπεδο διεθνές, μέσω του Συμβουλίου της Ευρώπης και μέσω των Ηνωμένων Εθνών, της πλατφόρμας του Πεκίνου, ε, μπορεί να υπάρχουν κάποιοι ε, μηχανισμοί παρακολούθησης, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να έχει και δικούς της μηχανισμούς. Ε, τα κράτη-μέλη μπορούν να δεσμευθούν μέσα στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Μπορούμε να τα πετύχουμε όλα αυτά. Αν έχουμε αποτελεσματική εφαρμογή και διαδικασία παρακολούθησης, μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι οι δεσμεύσεις επιτυγχάνονται. Και όταν δεν επιτυγχάνονται, μπορούμε να θέσουμε ερωτήματα. Γιατί συνέβη αυτό, τι μπορούμε να κάνουμε. Χωρίς όλα αυτά, χωρίς όλες αυτές τις δεσμεύσεις, είναι δύσκολο να δούμε πώς τα επόμενα 5, 10, 20 χρόνια θα έχουμε πραγματική αλλαγή σε, μια, σε έναν τομέα ο οποίος χρειάζεται όχι μόνο άμεσες ε, λύσεις, αλλά και μακροπρόθεσμες ε, ε, λύσεις σε επίπεδο πολιτιστικό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Λέβεν. Νομίζω ότι στην παρουσίασή σας θέσατε πολύ σημαντικά ζητήματα. Τα έχουμε συζητήσει επανειλημμένως στη δική μας Κοινοβουλευτική Επιτροπή και πολύ σωστά λέτε ότι το πρόβλημα είναι διαρθρωτικό, δομικό. Ξεκινούμε από μια άνηση κοινωνία και η ανισότητα των δύο φύλων δημιουργεί τέτοιου είδους καταστάσεις, όπως είναι η καταπολέμηση της βίας ενάντια στις γυναίκες. Πρέπει λοιπόν να δουλέψουμε με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, να έχουμε μια πιο ίση κοινωνία, να αξιοποιήσουμε την εκπαίδευση, την παιδεία, να επιφέρουμε τις απαραίτητες θεσμικές αλλαγές και πρέπει να δουλέψουμε και πιο βραχυπρόθεσμα με πιο συγκεκριμένες πολιτικές όπως είναι η αντιμετώπιση των θυμάτων βίας, να δουλέψουμε καλύτερα στο δικαστικό και αστυνομικό κομμάτι. Θέσατε λοιπόν επιτάπητος αυτά τα ζητήματα και υπογραμμίσατε κάτι που εμείς ως Επιτροπή ε, ενστερνιζόμαστε και έχουμε διεκδικήσει επισταμένως. Δηλαδή ότι είναι ανάγκη να έχουμε ομοιογενή, ομοιόμορφα στατιστικά στοιχεία, έγκυρα, για να μπορούμε να έχουμε εργαλεία πάνω στα οποία θα στηριζόμαστε, να μπορούμε να τα εφαρμόσουμε σε διάφορους τομείς. Αυτό το απαιτούμε. Ανέκαθεν το έχουμε απαιτήσει. Είναι ένα έργο απαραίτητο και ελπίζω να αναλάβουν οι θύνοντες και την απαραίτητη πολιτική ευθύνη για να το φέρουν σε πέρας. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβασή σας. Υπάρχουν ερωτήσεις, θα ήθελε κάποιος ή κάποια να θέσει κάποιο θέμα στον κύριο Λέβεν. Έχουμε λίγο χρόνο. Ναι, παρακαλώ εσείς να μας πείτε πρώτα το όνομά σας και να μην μακρηγορήσετε. Η ερώτηση είναι σύντομη για να ακούσουμε και τους υπόλοιπους και να συνεχίσουμε και την ημερήσια διάταξη, την εξέτασή της. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σας. Λέγομαι Αντώνιο Σύντορα και είμαι σύμβουλο σε θέματα φίλων, δύο φίλων. Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Σε αυτό το έργο έγκρισης κριτηρίων, ομοιόμορφων κριτηρίων ώστε να εκπονηθεί γενική στρατηγική, ποιοι είναι οι πιο έγκυροι δείκτες ποια είναι τα κριτήρια τα οποία οπωσδήποτε πρέπει να είναι παρόντα και δεν επιτρέπεται να απουσιάσουν από μια γενική στρατηγική. Είναι ένα ολόκληρο ζήτημα το όλο θέμα, η όλη συζήτηση για τους δείκτες, αλλά ποια είναι, εν πάση περιπτώσει, τα χαρακτηριστικά των δικτών ε, που τους καθιστούν ως τους πλέον, πλέον κατάλληλους για, ε, για τη χάραξη ευρύτερης γενικής στρατηγικής. Ευχαριστώ. Απάντηση. Δεν ξέρω ε, εάν θα αναπτυχθούν ε, δείκτες μέσα σε μία και ενιαία στρατηγική. Δεν ξέρω αν αυτό είναι το θέμα και το ζητούμενο. Δεν πετυχαίνουμε έτσι πάντοτε τους στόχους μας. Ε, ωστόσο, ένας απλός δείκτης ή και στόχος είναι π.χ. ο αριθμός των γυναικών που αναφέρουν ότι έχουν υποστηβία, ότι έχουν υπάρξει θύμα βίας αυτό θα είναι καθεαυτό δύσκολο. Και από εκεί και πέρα αποφασίζει, αποφασίζει κανείς αν θα δώσει σημασία στο είδος του αδικήματος που διαπράτεται, στις αναφορές που υποβάλλονται ή σε κάποιο άλλο σκέλος αυτού του προβλήματος. Το ΦΡΑ, η Υπηρεσία για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα, έχει ήδη εδρεώσει ένα τρόπο έβρεσης ε, των πληθυσμών στόχων. Εάν ε, πάρουμε αυτό τον τρόπο εργασίας και εστιάζουμε την προσοχή στους δύο-τρεις βασικούς δείκτες που το ΦΡΑ, η υπηρεσία αυτή, έχει ε, υιοθετήσει, τότε μπορούμε να έχουμε αποτελέσματα. Το σημαντικό είναι να ε, έχει κανείς έναν π.χ. στόχο και να δει πώς εξελίσσεται αυτό, σε ποια, πώς αλλάζουν τα νούμερα σε βάθος χρόνου. Σήμερα δεν μπορούμε να ξέρουμε αν οι πολιτικές είναι επιτυχημένες γιατί δεν ξέρουμε το σημείο κίνηση με τι νούμερα ξεκινήσαμε, με πόσους ανθρώπους. Το επίπεδο της βίας είναι κομμάτι λοιπόν αυτού του παζλ. Άλλο κομμάτι είναι ο βαθμός στον οποίο ε, παίρνουν το λόγο δημόσια οι γυναίκες, δηλαδή αναφέρουν αυτό το οποίο έπαθαν, άρα τα στατιστικά στοιχεία των αδικημάτων. Και ε, τρίτος στόχος ή δείκτης μπορεί να είναι ο δείκτης ανταπόκρισης και προστασίας που σε πόσες περιπτώσεις ήρθαμε ε, και παρήχαμε στήριξη ή προστασία. Αυτά τα τρία νούμερα λοιπόν θα μπορούσαν να είναι χρήσιμοι δείκτες. Π.χ. έτσι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε στο πόσα καταφύγια ε, και καταλήμματα θα πρέπει να υπάρχουν στα κρατη και χρειάζονται τα κρατη με τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης ξέρουμε πώς θα προσεγγίσουμε τη στρατηγική. Το θέμα είναι να εστιάσουμε την προσοχή μας σε κάθε ένα από αυτά τα σκέλη. Η Πρόεδρο, σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά τον κύριο Λέβεν για τη συνεισφορά του. Είναι πολύ σημαντική για τις συζητήσεις που θα έχουμε τους επόμενους μήνες στην κοινοβουλευτική μας επιτροπή. Ελπίζω να μπορέσουμε να συνεργαστούμε ξανά μαζί του στο μέλλον, να είναι σε θέση να συνεχίσει να συνεισφέρει στη δουλειά μας και μάλιστα το συντομότερο δυνατό και ελπίζω το συντομότερο δυνατό με το νομοθετικό έργο των ε, ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων να εξαλειφθεί το γρηγορότερο ε, αυτή η μάστιγα της βίας κατά των γυναικών έτσι ώστε να προχωρήσουμε τελικά σε μια πιο ίση και δίκαιη κοινωνία. Αν συμφωνείτε να περάσουμε στην τελευταία παρέμβαση του εργαστηρίου μας, στο τελευταίο σημείο, μάλλον, πολιτικές της ισότητας των φύλων στο πλαίσιο της ε, διεθνούς πολιτικής εξωτερικών υποθέσεων και της αναπτυξιακής πολιτικής. Όλα αυτά είναι σημαντικά. Είναι στην ημερήσια διάταξη, στο πρόγραμμα εργασιών της Επιτροπής αυτής. Έχουμε εκθέσεις όπως αυτή για την αξιολόγηση και για την κατάσταση της πλατφόρμας του Πεκίνου, ε, την ε, εξέταση των στόχων της χιλιετίας υπό το πρίσμα της ισότητας των φύλων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας παίκτη καθοριστικός ε, στην ε, διεθνή πολιτική και η πολιτική συνεργασίας και ανάπτυξη στην οποία χαράσει η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να οδηγήσει στην εξάλληψη ή στην άμβληση, εν πάση περιπτώσει, των ανισοτήτων μεταξύ των δύο φύλων και σε άλλες περιοχές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δίνω το λόγο στην κυρία Πέτρα Ντεμπούσνερ από το Πανεπιστήμιο της Ανβέρσας του Βελγίου. Σας ευχαριστώ θερμά που ήρθατε. Είστε εδώ μαζί μας με όλες εμάς και όλους εμάς και θα σας ε, δώσω το λόγο για να μιλήσετε για όλα αυτά τα θέματα που μόλις τώρα ε, παρουσίασα και αν έχουμε χρόνο στη συνέχεια θα κάνουμε και συζήτηση. Σας ευχαριστώ πολύ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Δεν έχουμε πολύ χρόνο και γι' αυτό δεν θα σας παρουσιάσω το πίνακα με τα, το πίνακα SWOT με τα ισχυρά σημεία και τα αδύνατα σημεία, τους κινδύνους και τις ευκαιρίες. Θα σας παρουσιάσω τα συστάσεις, γιατί αυτό είναι και το πιο χρήσιμο για εσάς. Αυτό το οποίο χρειάζεται λοιπόν, ε, γιατί στρατηγική της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών 2016-2020 είναι η βελτίωση του συντονισμού ε, των, δράσ, ε, ε, των υπηρεσιών εξωτερικής δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να καταλήξουμε σε μια νέα στρατηγική ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών για το 2016 μέχρι και το 2020. Πρέπει να υπάρχει συνέπεια στην πολιτική. Άρα η κάθε γενική διεύθυνση η οποία είναι αρμόδια, η γενική διεύθυνση για την την εξωτερική πολιτική, η υπηρεσία εξωτερική δράση, η Γενική Διεύθυνση για την Ανάπτυξη, για τη διεύρυνση, για το εμπόριο. Πρέπει όλε αυτέ οι γενικέ διευθύνσει να επιφορτιστούν με νέα καθήκοντα, με νέε ευθύνε. Π.χ. η Γενική Διεύθυνση Trade για το διεθνέ Εμπόριο απουσιάζει παντελώ Η Γενική Διεύθυνση για τη Διεύρυνση είναι παρούσα, αλλά α το πούμε με ειλικρίνεια. Οι στόχοι που έχει θέσει δεν είναι καθόλου φιλόδοξοι. Ένας από τους στόχους της είναι να παρακολουθεί ε, την εφαρμογή και την στήριξη και την προσχώρηση στα κριτήρια της Κοπενχάγης. Πολύ ωραία διατύπωση, αλλά εξαιρετικά ασαφής, ευρεία και είναι εξαιρετικά δύσκολο να το παρακολουθήσει αυτός. Κανείς αυτό κάθε χρόνο μπορεί να δώσει δύο-τρία παραδείγματα και έτσι να συντάξει μια πολύ όμορφη έκθεση, αλλά δεν ε, εντάσει τη διάσταση του φύλου με συστηματικό τρόπο σε όλες τις πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης με αυτόν τον τρόπο. Το σημαντικό είναι να είναι όλοι στο τρένο, αν θέλετε, να μην μείνει κανείς εκτός από όλες αυτές τις γενικές διευθύνσεις. Και κάθε τέτοια υπηρεσία θα πρέπει να έχει καταρτήσει εσωτερικό σχέδιο δράσης για το πώς θα κάνει συστηματικά gender mainstreaming, στις διάφορες ε, πολιτικές και θα πρέπει να περιλαμβάνει και όλες τις πτυχές αυτών των πολιτικών. Άρα, οι γενικές διευθύνσεις για το διεθνές εμπόριο, για τη διεύρυνση, αλλά και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την εξωτερική δράση πρέπει να ξεκινήσουν ήδη την κατάρτιση αυτού του εσωτερικού σχεδίου δράσης, να προβούν σε ανταλλαγή καλών πρακτικών ε, που ε, έχουν ήδη οι γενικές διευθύνσεις για, ε, για την ανθρωπιστική βοήθεια ΕΚΟ και ΑΦΚΟ. ένα συνολικό σχέδιο θα ωφελήσει όλους τους ε, παίκτες έτσι ώστε όλοι να ενταχθούν και να εμπλακούν σε αυτή την προσπάθεια. Οι διάφορες γενικές διευθύνσεις μπορούν να διδάξουν η μία την άλλη, να, μοιραστούν η μία με την άλλη τις καλές ε, πρακτικές. Η τέφκο για παράδειγμα για την αναπτυξιακή συνεργασία μπορεί να ε, μεταφέρει στις υπόλοιπες γενικές διευθύνσεις τους ε, σχετικούς δείκτες, τους πολύ χρήσιμους του ε, ΟΣΑ. Και θα μπορούσε ενδεχομένως να ενημερώσει για θέματα εμπορικής πολιτικής. Αξίζει να διερευνηθούν αυτές οι οδοί Gender, Focal Persons Network, δηλαδή ένα δίκτυο των συνδέσμων οι οποίοι είναι κυρίως επιφαρτισμένοι με την παρακολούθηση των θεμάτων που έχουν να κάνουν με τη διάσταση των φύλων, του φύλου ε, στις χώρες αυτές. Αυτό θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμο. Σε γενικές γραμμές, η πολιτική για τα φύλλα πρέπει να διευρυνθεί και να εμβαθυνθεί, να ισχύσει και να εφαρμοστεί περισσότερο στις εξωτερικές σχέσεις και στην αναπτυξιακή βοήθεια που δίδουμε. Ε, συντάσσονται πάρα πολλές εκθέσεις, υπάρχει ένα momentum, μια όθηση δηλαδή για όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία εξελίσσονται, αλλά να γνωρίζουμε και την αφήγηση η οποία έχει την προτίμηση των περισσότερων αυτή τη στιγμή. Η τάση είναι να μην ανοιχνεύεται η πρόοδος. Τι γίνεται σε όλες αυτές τις εκθέσεις των ειδικών, των εμπειρογνωμόνων, των διαφόρων, παρουσιάζουν ε, ε, συγκεκριμένα γεγονότα τυχεοποιημένα αν θέλετε, δεν παρακολουθούν προοδευτικά σταθερά ακριβώς τι γίνεται και καλό θα ήταν να μπορούμε να συγκρίνουμε τους, τις εκθέσεις ετησίως σε κάθε χρόνο. Τώρα, ως προς τα πλεονεκτήματα του προηγούμενου πλαισίου για τους στόχους της χιλιετίας, ε, πλέον οι στόχοι είναι πολύ πιο απτοί. Ωστόσο, είναι στόχοι εφαρμοστικοί για να είναι απλοί. Δεν είναι ιδιαίτερα στόχοι που θα αλλάξουν εκ βάθρων μια κατάσταση. Π.χ. Ε, η ενδυνάμωση οικονομική των γυναικών, η συμμετοχή τους στην πολιτική ζωή, στη στρατηγική μετά το 2015. Όλα αυτά είναι πιο θεωρητικοί, πιο γενικοί στόχοι και πρέπει να έχουν πιο λεπτομερείς δείκτες ε, που θα τους αξιολογούν. Η πρόσβαση σε μια αξιοπρεπή εργασία, ε, η πρόσβαση σε δίκτυο, σε οτιδήποτε. Γενικά το gender mainstreaming πρέπει να σας πω ότι δεν είναι ε, στρατηγική χωρίς καθόλου κόστος ή ελάχιστο κόστος. Είναι στρατηγική που έχει κόστος και άρα θα πρέπει να αυξηθούν οι πόροι, ώστε να εφαρμοστούν συγκεκριμένα έργα, να γίνουν συγκεκριμένα έργα για το empowerment των γυναικών, να αποκτήσουν δηλαδή ε, δύναμη αν θέλετε, να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους. Και οι πόροι αυτοί πρέπει να γίνεται παρακολούθησή τους, του τρόπου με τον οποίο αξιοποιούνται και χρησιμοποιούνται σε βάθος χρόνου. Εγώ έχω ασχοληθεί με αυτό τα τελευταία χρόνια. Ανοιχνεύω, εντοπίζω πόσα χρήματα πάνε στο gender mainstreaming, πόσα πάνε σε συγκεκριμένα έργα, πόσα πάνε σε οργανώσεις γυναικών και είναι ένα ε, ε, καθήκον σχεδόν ανέφικτο, αδύνατο να υλοποιηθεί. Απλά δεν υπάρχουν στοιχεία. Και να ενταχθεί αυτό στην αιτήσια... Ε, έκθεση των γενικών διευθύνσεων και σίγουρα η Γενική Διεύθυνση για την Αναπτυξιακή Συνεργασία και Βοήθεια, η ΔΕΦΚΟ, πρέπει στην ετήσια έκθεση απολογισμού της κάθε χρόνο να περιλαμβάνει συγκεκριμένο κεφάλαιο για αυτό το θέμα. Δεν το κάνει τώρα, δεν γίνεται τώρα, δεν υπήρχε στην τελευταία έκθεσή της. Και νομίζω ότι εσείς ως Επιτροπή του και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις γυναίκες πρέπει να το παρακολουθήσετε στενά το ζήτημα αυτό. Άλλη σύσταση τώρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πρωτοπόρος στην αξιοποίηση εργαλείων του προϋπολογισμού για την επίτευξη αυτών των σκοπών. Άρα, στις ε, εφαρμοστικές λεπτομέρειες θα πρέπει να περιγράφονται και οι στόχοι που έχουν να κάνουν με τα δύο φύλλα. Δηλαδή, στηριζόμαστε όλο και περισσότερο στον προϋπολογισμό για να πετύχουμε αυτούς τους στόχους, αλλά δεν, δεν έχουμε ε, ιδέα περί του τι ακριβώς συμβαίνει στην πράξη, ποιες είναι αυτές οι οκτώ εφαρμοστικές λεπτομέρειες, γιατί ο δείκτης του ΩΣΑ δεν περιλαμβάνει το budget support, τη στήριξη από τον προϋπολογισμό. Και ε, στο 90% των περιπτώσεων οι στόχοι ή οι δείκτες των δύο φύλων δεν είχαν συμπεριληφθεί στα ε, διαρθρωτικά ή γενικά προγράμματα για τη στήριξη του προϋπολογισμού. Ενώ όταν μίλησα με τα αρμόδια στελέχη, μου είπαν ότι αυτό είναι μια εξαιρετική δικαιολογία με την έννοια ότι είπαν ότι εγώ για παράδειγμα για τον εαυτό τους δεν ε, ε, κάνω έργα, εγώ κάνω budget support. Δεν πρόκειται να βγάλω αυτό το δίκτυο από το συνολικό άθροισμα έτσι ώστε να φανεί η διαφορά της διάστασης του φύλου γιατί είναι τόσο λίγοι οι δείκτες που δεν αξίζει αυτό, θα χάσουμε και τη γενικότερη εικόνα. Τα λέω όλα αυτά για να σας δείξω ότι ε, όσοι δουλεύουν επί τόπου δεν έχουν ιδέα για αυτά τα ζητήματα. Ξέρω ότι η Γενική Διεύθυνση DEFCO έχει κάνει εκπαίδευση για το budget support. Ε, αν όμως δεν δοθούν κίνητρα και πρωτοβουλίες δεν αναλυθούν, δεν θα γίνουν και πολλά πράγματα. Και υπό αυτή την έννοια καλό είναι να πω ότι έχουμε πράγματι πάρα πολύ καλές βέλτιστες πρακτικές. Π.χ. η μελέτη UNIFAM της Επιτροπής, όπου τα θέματα τα οικονομικά και του προϋπολογισμού έχουν ενταχθεί στη διαμόρφωση της ημερήσιας διάταξης και ε, φαίνεται ξεκάθαρο πώς έχουμε αποτέλεσμα στην πράξη. Υπό μια πολύ καλή πρακτική στο Μαρόκο, για παράδειγμα, που αξίζει τον κόπο να διαδοθεί. Όμως όλα αυτά δεν έχουν βρει τη θέση που τους ταιριάζουν στην ευρύτερη ε, συνεργασία ε, στο εσωτερικό της, ε, των φορέων των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, Χρειαζόμαστε πιο ισχυρή πολιτική ηγεσία, μεγαλύτερη πολιτική βούληση και λογοδοσία των ανώτατων στελεχών στην περιγραφή για την εκάστοτε θέση, στην αξιολόγηση των επιδόσεων ε, ανωτέρων και ανωτάτων στελεχών, θα πρέπει να ε, είναι προαπαιτούμενο να έχει κάποιος μια κάποια ειδίκευση, μια κάποια γνώση και μάλιστα επαρκή των διαστάσεων του ε, φύλου. είναι μια βασική ε, αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις περιπτωσιολογικές μελέτες που έχω κάνει κάθε φορά είδα και έχει αποδειχθεί ότι κάθε φορά που ο επικεφαλής μιας αντιπροσωπείας ή ο επικεφαλής ενός τμήματος αν θέλετε έχει ο ίδιος ενεργά ασχοληθεί με το gender mainstreaming τότε αυτό κινητοποιεί όλη την ομάδα των υφισταμένων του και τα αποτελέσματα είναι πολλαπλάσια. και βέβαια στο πολιτικό διάλογο με τις τρίτες χώρες για το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το θέμα της προσχώρησης, ε, για το διεθνές εμπόριο και ούτω καθεξής, υποτίθεται θεωρητικά πάντοτε ε, υπάρχει και το, η διάσταση του φύλου, αλλά στην πράξη δεν δίνουμε τόσο μεγάλη σημασία. Στην Αφρική, για παράδειγμα, δεν θεωρείται θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων η βία με βάση το φύλλο λόγω της κατάστασης. Σημαντικό είναι λοιπόν να ενημερώνουμε και να εκπαιδεύουμε τους δικούς μας ανθρώπους που στέλνουμε ως συνομιλητές σε τέτοιου είδους συζητήσεις. Και τέλος, το προσωπικό ε, που ασχολείται με την εξωτερική δράση ε, η υφίσταται εκπαίδευση από την ΤΕΦΚΟ, αυτό ισχύει μεν, αλλά αν δεν του δοθούν περαιτέρω κίνητρα αν δεν κινητοποιηθεί περαιτέρω, δεν ε, έχουμε αποτελέσματα. Να, νομίζω ότι για ορισμένα στελέχη, ορισμένες κατηγορίες της διοίκησης θα πρέπει να είναι υποχρεωτικό όσοι ασχολούνται με τα εξωτερικά να ακολουθήσουν το training και τις ε, εκπαιδεύσει που προσφέρει η DEFCO. Και τέλος, τα gender focal persons και στα κεντρικά, τα αρχηγεία και στις αντιπροσωπείες. Οι άνθρωποι δηλαδή που ασχολούνται με, κυρίως και δίνουν έμφαση στη διάσταση του φύλου. Θα πρέπει να μπορούν να, όλο το ωράριό τους να το αφιερώνουν σε αυτό το θέμα και να ε, προσληφθούν ε, περαιτέρω εμπειρογνώμονες σε ανώτερα επίπεδα της διοίκησης για να μην ε, ε, χαθεί ο πλούτος τους όταν αποσπώνται και μετατίθενται αλλού, να υπάρχει συνέχεια στη γνώση και σε όλη αυτή τη δουλειά που έχουν αποκομίσει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Προεδρεύουσα. Είναι σημαντικές ενδιαφέρουσες θέσεις ε, οι θέσεις σας γιατί βλέπα, είδαμε αυτά τα κενά αυτά τα θέματα που εδώ στην Επιτροπή και από την εργασία μας σαν βουλευτές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σε σχέση με την ε, Επιτροπή και στις διάφορες γενικές διευθύνσεις στην εργασία. Όλα αυτά θα μπορούσαν να είναι κάτι το σημαντικό. Γιατί είδαμε, θίξατε αυτά τα κενά, μιλήσαμε και εμείς για αυτά, για την ανάγκη μιας εκπαίδευσης, μιας όθησης. Ε, επιμένω ότι πραγματικά ήταν κάτι το πολύ σημαντικό. Ξεκινάμε τώρα τις παρεμβάσεις, να ακούσουμε τα σχόλια, ορισμένε ερωτήσει σχετικά. Η συνάδελφος συζήτησε το λόγο. Ναι, ναι. Θα μιλήσω και εγώ για σε ισπανικά αν θέλετε. Ευχαριστώ. Εργάζομαι σε εξωτερικές υποθέσεις παρά στις γυναίκες Αυτά που ακούσαμε ήταν πολύ ενδιαφέροντα από την κυρία Ντεμπούσερ. Θα πρέπει να δούμε την κατάσταση που αντιμετωπίζουμε με την Επιτροπή. Θα πρέπει να δούμε πώς γυναίκες θα είναι εδώ. Και είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Δεν ξέρω, θα φτάσουμε το 40% που ζητήσαμε. Τα κράτη-μέλη προσπαθούν ώστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτό που είχε ζητήσει και το 2012 σχετικά με την έκθεση Καϊτεκάινεν ε, να υπάρχει ένας άνδρας μία γυναίκα. Δεν ξέρω, νομίζω ότι σε αυτά τα πλαίσια λοιπόν βρισκόμαστε και δεν μας εκπλήσει ότι εξακολουθούμε να λειτουργούμε με τον τρόπο αυτό, τα πράγματα δεν πάνε όπως πρέπει. Διάφορα σχόλια Εγώ προσέξα αυτό που είπε η κυρία Ντεμπούσερ. Στο τις εκθέσεις μας και στην ε, Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων ήμουν για το 25 εγώ τα τελευταία πέντε χρόνια. Σε κάθε μία από τις εκθέσεις και της Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πάντα περιλαμβάνεται και μία παράγραφος για τις ευκαιρίες, για την κατάσταση στις γυναίκες αλλά αυτά είναι ορισμένα σημειακά στοιχεία. Αυτό συνέβη εδώ, αυτό συνέβη εκεί. Δεν είναι όμως κάτι το γενικό. Θα πρέπει να δούμε, να ελέγξουμε σε σχέση με πέρυσι, με πρόπερση, η κατάσταση πώς εξελίσσεται. Θα πρέπει αυτό να γίνει κατά συστηματικό τρόπο και στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εντάξει, σχόλιο είναι, δεν είναι ερώτηση. Μια ερώτηση, ναι, ίσως. Δεν πρέπει να έχει να κάνει μόνο με την ανάπτυξη της εξωτερικής υποθέσεως, αλλά κάτι το γενικότερο. Αλλά και με άλλους που είναι εδώ παρόντες. Από τη στιγμή που μιλάμε για στρατηγικές πριν να είμαι βουλευτής εργάστηκα σε θέματα βίας κατά των γυναικών. Πολύ σημαντικό είναι να υπάρξουν άνδρες που να ενημερωθούν σχετικά. Δεν ξέρω πώς το λένε στα ισπανικά, είναι αυτή η εκστρατεία του White Ribbon που λέει ότι υπάρχουν διάφοροι που λένε ότι είναι κατά της βίας ε, στις γυναίκες. Θα πρέπει να διεξαχθεί αυτή η μάχη και από άντρες, γυναίκες με τους συντρόφους της. Είναι σημαντικό. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε χωρίς την εργασία των ανδρών. Δεν μπορεί να επιτευχθεί αυτό με νόμους και μόνο. Είναι θέμα της ίδιας κοινωνίας. Ένα ερώτημα. Μήπως θα μπορούσατε να μας επαναλάβετε μια έκθεση είπατε για μια-δυο χώρες όπου υπήρξαν σημαντικά παραδείγματα. Το Περού νομίζω μια άλλη χώρα δεν την άκουσα. Γιατί νομίζω ότι τα παραδείγματα θα μπορούσαν να δείξουν τι πρόοδος έχει επιτευχθεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία μου σε σχέση με το θέμα που αναφερθήκατε για τη σύνθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αύριο είπαμε ότι θα στον κύριο Γιούνκερ σαν πρώτης επιτροπής θα θίξουμε αυτή τη θέση μας, ότι την προβάλλουμε και θα πρέπει να υπάρχει μια ισορροπημένη ισχυρή εκπροσώπηση των γυναικών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας είπαν ότι μέχρι σήμερα θα είχαμε 7 υποψήφιες γυναίκες σαν επιτροπή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι παρακάτω χαμηλότερο αριθμό από το σημερινό. Δεν ξέρω, δεν, ξέρω, δεν νομίζω να προχωρήσω. Δεν έχουν προχωρήσει αυτά τα χρόνια. Αντίθετα πήγαμε πίσω. Θα επαναλάβουμε τη θέση εδώ Επιτροπής, θα την επαναλάβουμε και πάλι στον κύριο Γιούνκερ. Ελπίζω δε ότι θα υπάρξουν τις επόμενες μέρες ή εβδομάδες παρόμοιες κινήσεις. Διαφορετικά θα δώσουμε άσχημο παράδειγμα από εδώ. Ακριβώς ε, ζητάμε μια κοινωνία με ίση εκπροσώπηση και το 50% των κατοίκων είμαστε γυναίκες αλλά στα εδώ όπου λαμβάνονται πολιτικές σημαντικές αποφάσεις για τις ζωές μας είμαστε υποεκπροσωπούμενες ε, θα πρέπει να το απαιτήσουμε αυτό και από το Κοινοβούλιο και έχετε το λόγο κυρία Ντεμπουσέρ για να απαντήσετε στο θέμα αυτό που αναφέρθηκε η προηγούμενη ερωτούσα. Ευχαριστώ. Thank you uh, for your Ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Δυστυχώς, ε, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να συμφωνήσω με αυτά που λέτε, ότι χρειαζόμαστε περισσότερους άντρες μαζί μας και αυτό που έχουμε δει στις ε, αντιπροσωπείες είναι ότι δεν έχει σημασία εάν είναι άνδρες ή γυναίκες ε, για να αλλάξουν πολιτικές. Το θέμα είναι πώς φτάνουμε εκεί. Φυσικά η πολιτική διοίκηση και η λογοδοσία των ανώτατων διοικητικών στελεχών είναι σημαντικό. Ε, χρειάζεται υποχρεωτικά κατάρτιση. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι συντάσσονται, αλλά τουλάχιστον έχουμε τη γνώση. Επίσης συμφωνώ ότι χρειαζόμαστε περισσότερους άντρες να εμπλακούν σε αυτόν τον πόλεμο για την ισότητα των φύλων και η πολιτική είναι ένας χώρος που κυρίως υπάρχουν ε, άντρες, όμως τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι αλλάζουν τα πράγματα και αυτό ε, επηρεάζει νομίζω και τις πολιτικές επίσης. Το ΙΕΣ έχει ε, κάνει κάποια πράγματα για να αλλάξει αυτό και παρόλο που χρειαζόμαστε τους άντρες μαζί μας, χρειαζόμαστε και γυναίκες σε υψηλές θέσεις να αποτελούν παράδειγμα γιατί έτσι θα αλλάξουν ε, και οι νοοτροπίες των αντρών. Επίσης υπάρχει μια μελέτη της Επιτροπής UNIFAM η οποία ε, βγήκε το 2008 και αναφέρεται σε χώρες στις οποίες υπήρχε υποστήριξη μέσω του προϋπολογισμού για να μπορεί κανείς να ευαισθητοποιηθεί στο θέμα της ισότητας των φύλων και είχαμε θετικές εξελίξεις. Γιατί είναι τόσο θετικές, γιατί η υποστήριξη του προϋπολογισμού είναι μια τεράστια ευκαιρία για την ισότητα των φύλων. Δεν είναι μόνο μια παγίδα όπως ήταν ως τώρα. Γιατί πρέπει να αναδιατυπώσεις τις δομές, να δεις τη διακυβέρνηση, Υπάρχει δηλαδή μια τεράστια ευκαιρία το περιεχόμενο να δίνει περισσότερη σημασία στην ισότητα των φύλων, να ενσωματώνεται η διάσταση του φύλου και σε επίπεδο περιεχομένου, αλλά και ε, ως προς το ότι έρχονται περισσότερες γυναίκες στο προσκήνιο. Αυτές βέβαια οι βέλτιστες πρακτικές δεν έχουν μπει στις ε, ευρύτερε πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υποστήριξη του προϋπολογισμού και πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επαναδεσμευτεί για αυτή την υποστήριξη. Αλλά αυτό που είδα είναι ότι τώρα υπάρχει λιγότερη διάσταση του φύλου στις ε, γραμμέ και τις εφαρμοστικές κατευθυντήριες γραμμές από ό,τι υπήρχε παλιά. Αυτό είναι ανησυχητικό γιατί χάνεται μια ευκαιρία. Πολύ καλά. Τελειώσαμε λοιπόν με το σημείο αυτό και θα ήθελα να επαναλάβω τις ευχαριστίες μας ε, τις συναδέλφους που με τις ερωτήσεις τους εμπλούτησαν ε, τη συζήτηση για θέματα που επαναλαμβάνω θα είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά για την εργασία της Επιτροπής μας και την κοινοβουλευτική μας εργασία, την προσεχή τους επόμενους μήνες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για τις εισηγήσεις ε, όσες συμμετείχαν σε αυτή την εργασία, σε αυτό το workshop. Σας ευχαριστούμε πραγματικά.